Thank you, for being... Καλημέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε αγαπητοί φίλοι. Ξεκινάμε αμέσως με το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ελπίζω όλοι σας να θα θελήσετε να συμμετάσχετε στην αντική συζήτηση Στον κύριο Μπάλλας θα δώσουμε πρώτα το λόγο, που είναι εισηγητής για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από όταν επιφορτίστηκα με αυτή την έκθεση, ήθελα να συναντήσω τους διάφορους συνομιλητές μου. Πήγα στη Βαρσοβία καταρχάς να συζητήσω με τις αρχές με την πολωνική κυβέρνηση, τα συνδικάτα, τους εκπροσώπους των επιχειρηματιών. Το ίδιο έκανα και στο Βερολίνο. Ακολούθησα το ίδιο σχήμα και συζήτησα με πολλούς ε, εκπροσώπους της κυβερνήσεως αλλά και με ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες, με εκπροσώπους των επιχειρηματιών και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο μετά συνέταξα αυτή την πρώτη πρόταση εκθέσεως που θα σας παρουσιάσω. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες με τους κοιόδης ηγητές. Και αυτό που εφαρμόζω και θέλω είναι να συναντώ τους κοιόδης ηγητές έναν έναν αρχικά για να γνωρίσω τις πρώτες τους εντυπώσεις και μετά ξεκινάμε τις πρώτες συνεδριάσεις όλοι μαζί για να δούμε όσο πιο γρήγορα να προχωρήσουμε, ξέροντας ότι στο, ποιος είναι ο ρυθμός των εργασιών ε, στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο ο ρυθμός των Υπουργών μας απασχολεί. Το, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ετοίμα το κείμενο για τη διευκόλυνση τη μετακίνηση των εργαζομένων, χωρί να χάνουν τα δικαιώματά της στη μετακίνησή του. Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, την Νορβηγία και την Ελβετία και αυτό είναι εξασφαλίσουμε μια συνέχεια της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων όταν περνούν αυτοί οι άνθρωποι που μια εθνική δικαιοδοσία σε άλλη. άρα κινούμεθα εντός του συντονισμού και όχι εντός συναρμονίσεως. Κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, κάποιοι όχι, αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι ο συντονισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τροποποίηση όσον αφορά τον συντονισμό των ε, παροχών όσον αφορά την ανεργία, των επιδομάτων ανεργίας. Ε, για τους μισθωτούς, πολύ συχνά αυτή είναι η πρώτη στη έρευνα και ανησυχία, η ανεργία και τα επιδόματα ανεργίας. Όσον αφορά την αδυναμία εξαγωγή των παροχών την ανεργία, κάποιο που πάει να βρει απασχόληση στο εξωτερικό μπορεί να τηρήσει προσωρινά το δικαίωμα για το επίδομα ανεργία κατά τη διάρκεια διαμονή στο εξωτερικό. Αυτό επεκτείνεται από τρει μήνε στου έξι μήνε στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δυνατότητα τα κράτη-μέλη να επεκτείνουν την περίοδο. Δηλαδή κάθε χώρα μπορεί να φτάσει μέχρι τέλο όσον αφορά το επίδομα ανεργία αν το επιθυμεί. Κατά την άποψή μου, εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση σε αυτό το στάδιο και προτείνω ακόμα και επέκταση τη περίοδου εξαγωγή μέχρι το τέλος της θητείας της επιδόματος ανεργίας. Προβλέπει πιο μακρά περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέχρι να βρουν εργασία αυτοί που μετακινούνται. Συσχετίζουν την παράταση της διάρκειας του επιδόματος μέχρι ο άνθρωπος να μπορέσει να βρει μια απασχόληση. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος να χρησιμοποιήσει κανείς το επίδομα για να ψάξει να βρει δουλειά. Τώρα το, δεν είναι το ίδιο εξαγωγή των δικαιωμάτων με τον συμψηφισμό. Λοιπόν, θα πρέπει να βρει υπόψη την περίοδο ασφαλίσεως που έχει αλλού ο άνθρωπος όταν εργάζεται και σε αυτή τη χώρα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριμήνου. Αυτή είναι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Διαφορετικά, το κάτω μέλο που άσκησε την στεριότητά του προηγουμένω θα πρέπει να του καταβάλει τις, ε, τα επιδόματα ανεργία. Η παρούσα κατάσταση φαίνεται σχετικά συγχυχημένη για του αρμόδιου φορεί των κρατών μελών. Από την πλευρά μου, σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να επιμείνω επί το εξή. Δηλαδή, αυτό το άθισμα είναι η βασική αρχή τη ε, νομοθεσία. Όπω ε, το έδειξε και η μελέτη της Ευρωπα... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρουσιάστηκε χτε. Πέρα από τι διευκρινήσει που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, περιορίζει κάπω το πλαίσιο. Και γι' αυτό προτείνω να πάει σε ένα μήνα, κάτι που είναι αρκετό, η περίοδο ελάχιστα αστηριοτήτων πριν να γίνει ψηφισμό τη περίοδου των παροχών στη χώρα μέλος της τελευταίας δραστηριότητα. Δεν θα πρέπει να, περιορίζεται η μετακίνηση ε, του εργαζομένου από μέτρα ε, περιοριστικά όσον αφορά τα επιδόματα αυτά. Τρίτο θέμα. Να επιμείνω επ' αυτού. Δεν συζητείται εκτενώς, αλλά πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν σημαντικό. Δηλαδή των ε, μεθοριακών εργαζομένων πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το κράτος μέλος της τελευταίας απασχόλησης θα πρέπει να καταβάλει τα επιδόματα αναργία στου εργαζομένου σε παραμεθόρη περιοχή, εάν αυτοί άσκησαν μια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 12 μηνών. Αυτή είναι η δραστηριότητα. Κάτω από 12 μήνε, εκεί η χώρα διαμονή ασχολείται. Πέρα από του 12 μήνε είναι η χώρα που εργάζεται ο εργαζόμενο. Το κάτω μέλο διαμονή είναι αρμόδιο παρόλο που ίσως στη χώρα δραστηριότητα του καταβάλει τις εισφορές του. Εκείνοι που εισπράττουν τις εισφορές είναι επιφορτισμένες να δώσουν και τα επιδόματα ανεργίας θα πρέπει όμως να γίνουν και αναγκαίες διευκρινήσεις όσον αφορά διατάξεις, ούτως ώστε να αποφευθεί ότι αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην δημιουργήσει δυσκολίες σε πρακτικές, διοικητικές, γλωσσικές ή προσφοράς κατάρτισης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί η αρμοδιότητα της δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εξηγούμε εδώ. Σήμερα με αυτές προτάσεις κάποιος που εργάστηκε πάνω από 12 μήνες σε μια χώρα, ο οποίος είναι ανεργός, μπορεί να, μπορεί να θέλει να ψάξει να βρει δουλειά, γίνεται έλεγχο σε το πόσο ψάχνει να βρει ε, εργασία στη χώρα που εργάστηκε. Αν ζει σε άλλη χώρα, τι θα κάνει. Θα πρέπει να πηγαίνει τακτικά στις αρχές ανεργίας της χώρας όπου εργάστηκε, αλλά στην οποία δεν διαμένει και αυτό μπορεί να δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα αν δεν έχει αρκετούς πόρους, γλωσσικό πρόβλημα, διότι δεν μιλάει και τη γλώσσα και αν υπάρχει κάποια δικαστική διαφορά βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίων όπου δεν γνωρίζει τη γλώσσα αυτών, είναι πολύ δύσκολο για εκείνο να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Κατανοούμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, δεν πρόκειται περί αμφισβητήσεω τη. Απλώ θα πρέπει να δώσουμε τα μέσα τα κατάλληλα, ώστε να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των νικητικών αρχών και το βάρος το μέγιστο διοικητικό θα πρέπει να το η χώρα διαμονής και το ετούντος άσυλο. Άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα περίπλοκο, διότι το Συμβούλιο προχωρά αρκετά αργά όσον αφορά το ζήτημα, είναι το θέμα ειδικού κεφαλαίου όσον αφορά την περίθαψη μακράς διαρκείας ε, για τις ασθένειες, για την ασθένεια. Καταρχάς είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας, δηλαδή ένα ειδικό κεφάλαιο υπάρχει για τη θεραπεία μακράς περίοδου. Η Διοικητική Επιτροπή που είναι ένας φορέας που ασχολείται ακριβώς με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως πρέπει να συνεργαστεί πιο στενά με τους, εταίρους, με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτό το κεφάλαιο κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να μπορούν να, να παρουσιάζονται, υπάρχει επαφή με αυτού τους και να υπάρχει και εκπρόσωπος των, του ασθενούς ή των ασθενών και ο οργανισμός ασφάλισης να είναι παρόντος στην, στον καθορισμό των παροχών. Εκεί δεν θα πρέπει, πώς να το πω, να κάνουμε κάτι γραφειοκρατικό χωρίς να συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα ήταν κάτι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Η πρόταση έχει στόχο να λάβει υπόψη την πρόσφατη ε, το ΔΕΚ έχει δικαιοδοσία σε αυτή την πρόσβαση αυτών των ε, ανθρώπων που είναι κινητοί, ε, μετακινούνται μεν αλλά δεν είναι δραστήριοι οικονομικά να έχουν αυτέ τι παροχέ να καλύπτονται. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης ότι θα μπορεί να κωδικοποιήσει τις αποφάσεις που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σήμερα. Υπενθυμίζω ότι είμαστε νομοθέτες, γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει μεγάλο ρόλο νομολογία σήμερα, αλλά διότι πολύ συχνά δεν κάνουμε, δεν ασκούμε εμεί το ρόλο μας του νομοθέτου είτε το Συμβούλιο είτε εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι δικός μας ρόλος σήμερα να κωδικοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις παρόλο που προφανώς αυτή η νομολογία βαρύνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσει σε τυποποίηση των διαδικασιών που αφορούν την μορφή, τη χορήγηση και το περιεχόμενο των εγγράφων που πιστοποιούν ότι ανήκει κάποιο στο σύστημα κοινωνική ασφάλιση, ε, καθορίζονται οι όροι χορήγηση των εγγράφων και απόσυρση των εγγράφων όταν αμφισβητείται από κάποιο φορέα κράτου μέλου απασχόληση αυτά τα έγγραφα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων ε, διοικητικών φορέων. Η αρχή τη συνεργασία τη θεμητή θα πρέπει να καλύπτεται μέσω του ορισμού τη προθεσμία για απάντηση πολύ κρατάει περίοδο και αυτό εμποδίζει τι διάφορε δικήσει να κινηθούν σωστά και πιστεύω ότι η απουσία απάντηση κάτι που δεν είναι κανονικό, θα πρέπει να συμπιφέρει μια ε, μετακύληση των αρμοδιοτήτων. Αν δεν υπάρχει απάντηση από την αρμόδια αρχή όσον αφορά το έντυπο που αποδεικνύει ότι ανήκει κάποιο σε ένα σύστημα κοινωνική ασφάλιση, θα πρέπει τότε η αρχή, η ετούσα που είναι αρμόδια από εκείνη την στιγμή, δεν μπορεί να υπάρχει νομικό κενό και να επικρατεί η νομική αναρχία για να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των δικήσεων και εξασφαλίζεται η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Υποστηρίζω ότι ενός νέου κειμένου και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου που θα συνδέει τους διάφορους φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως όπως υπάρχει στο Βέλγιο βάσει του, του μοντέλου της, ε, να υπάρχει ηλεκτρονική κάρτα και να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής ασφάλειας. Και αυτές είναι, αυτές είναι προτάσεις που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν γέννη λοιπόν θα πρέπει ε, να γίνει εξυγχρονισμός ψηφιακός των ε, εγγράφων. Όταν πήγα στη Βαρσοβία και όταν πήγα στο Βερολίνο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν υπήρχε ομοφωνία τουλάχιστον επί ενός σημείου ήταν αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη να είμαστε μια ήπειρος όπου αυτού του είδους τα έγγραφα, αυτή η τεκμηρίωση δεν είναι ψηφιοποιημένη και αυτό δυσχεραίνει εξαιρετικά τους ελέγχους ε, φορτώνει τι επιχειρήσει, αυξάνει το διοικητικό του άχθο, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Θεωρώ σημαντικό να διευκρινίσουμε και του εφαρμοστέου κανόνε για του αποσπασμένου μισθωτού. Ελάχιστη υποχρεωτική περίοδο που ανήκουν στην κοινωνική προνοια του κράτου αποστολή. Θα πρέπει εκ των προτέρων να εκδίδονται τα διάφορα έγγραφα πριν την απόσπαση και για τους ανεξαρτήτους εργαζομένους και πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό και όσον αφορά τους ανθρώπους με πολλές δραστηριότητες. προτείνω επίσης μια τροπολογία των διατάξεων που προβλέπονται για να αποφευθεί ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει πρακτικέ δυσκολίε, διοικητικέ, γλωσσικέ ή προσφορά κατάρτιση και διευκρινιστούν οι αρμοδιότητε του δημόσιου τομέα και των διαφόρων φορέων των υπευθύνων για την απασχόληση όσον αφορά το θέμα των κοινωνικών εισφορών που πρέπει να καταβληθούν στην περίπτωση απόσπαση αλλά και των πολλαπλών δραστηριοτήτων. Προτείνω με την τροπολογία 54, δηλαδή ότι η αμοιβή όπω καθορίζεται αυτή μετά την αναθεώρηση τη οδηγία όσον αφορά του αποσπασμένου εργαζομένου αποτελεί τη βάση από την οποία οι κοινωνικέ εισφορέ υπολογίζονται. Δεν είναι ακριβές σήμερα, υπάρχουν κάποιες ερμηνείες ποικιλόμορφες Τροπολογία 25. Εγώ θα ήθελα επίσης να τροποποιήσω το άρθρο 16 που προβλέπει τώρα τα κράτη-μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν επί παρεκκλήσεων καθώς και αυτό το άρθρο χρησιμοποιείται για να επιτρέπει τώρα παρεκκλήσεις από την περίοδο των 24 μηνών που προβλέπεται για τη διάρκεια της απόσπασης. Παρομοίως, θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη όταν αυτό το επιθυμούν να καταρτήσουν μια κοινή, ένα κοινό καθεστώ κάλυψη κοινωνική για του αποσπασμένου εργαζομένου ε, και τα άτομα με πολλαπλέ δραστηριότητε, από τη στιγμή αυτό το καθεστώ κοινωνική προστασία να μην είναι πιο ευνοϊκό. Υπάρχει βασικό κανόνα, δηλαδή είναι ότι να ανήκει κάποιο στο σύστημα κοινωνική ασφάλιση σήμερα για του αποσπασμένου εργαζομένου, του ανεξαρτήτου ε, και του ανθρώπου με πολλέ δραστηριότητε. Θα πρέπει όμω μέσω διμερού συμφωνία να επιτρέπεται να προχωρήσει κανεί πιο μακριά, προφανώ σε ανώτερο επίπεδο και προστασία μεταξύ μεταξύ δύο χωρών που το επιθυμούν και έτσι να υπάρχουν κάποιοι πειραματισμοί που θα είναι χρησιμότατοι για όλου εν συνεχεία. Αν το αντικείμενο του κανονισμού είναι να υπάρχει συστονισμό των κοινωνικών συστημάτων, ε, δεν νομίζω να υπάρχει νομική αντίρρηση όσον αφορά την εναρμόνιση και ε, ομοιομορφία των συστημάτων κοινωνική ασφαλίσεω, αν το επιθυμούν αυτά τα κράτη-μέλη. Τέλο, είμαι αντίθετο ε, με ε, ε Να υπάρχει προσαρμογή για τα παιδιά. 1% των εισφορών πηγαίνουν στα παιδιά που ζουν σε άλλο κάτω μέλο από εκεί που εργάζονται οι γονεί. Και αυτό έχει αντίκτυπο στα δημοσιονομικά με ένα σύστημα προσαρμογή και χρειάζεται μια συνεχή επικαιροποίηση των, των ποσοστών αυτών, συναρτήση του τόπου διαμονή των παιδιών και είναι περίπλοκο το σύστημα αμφισβητήσιμο και εξαιρετικά γραφειοκρατικό και δεν βλέπω πώ σήμερα αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί πέρα από το θεωρητικό επίπεδο. Συμπέρασμα λοιπόν θα ήθελα οι συζητήσει όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για το συντονισμό να καταλήξει να, να μην καταλήξει σε κοινωνικό τουρισμό, απάτες και, και καλυμμένο προστατευτισμό. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Υπάρχουν κάποιες χώρες, βλέπετε, που έχουν την τάση να κατηγορούν άλλες χώρες ότι εφαρμόζουν τον κοινωνικό τουρισμό Δηλαδή, οι πίκοοι του κάνουν αυτό τον κοινωνικό τουρισμό. Είναι επιβλαβέ αυτό για αυτού που θέλουν να εργαστούν. Και από την άλλη πλευρά, πολύ συχνά θεσπίζουμε μέτρα τα οποία είναι μέτρα ελεγκτικά, ούτω ώστε να μην κάνει ο καθένα ό,τι θέλει και υπάρχουν κατηγορίε κοινωνικού προστατευτισμού. Α προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από αυτέ τι τοποθετήσει. Για μία ακόμη φορά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, αντιρρήσει ε, μεταξύ Βορρά και Νότου και διαφορέ μεταξύ Ανατολή και Δύση. Αυτό που υπάρχει σήμερα και ίσως να το οικοδομούμε αυτή την έκθεση, είναι η κινητικότητα των εργαζομένων που πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από όπου και αν προέρχονται και όπου και αν μεταβαίνουν. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό πνεύμα και σας ευχαριστώ πολύ. you for Ευχαριστώ για αυτά τα εισαγωγικά σας σχόλια, κύριε Μπαλάς. Τα μέλη της Επιτροπής σας παρακαλώ πολύ μην ξεπεράσετε τα δύο με 2,5 λεπτά όταν παίρνετε το λόγο. Για να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να υπάρξουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, εάν χρειαστεί. Ξεκινάω δίνοντας το λόγο στον κύριο Σούλτσε. Σας παρακαλώ πολύ, δύο με δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Κάποια πάρα πολύ θετικά στοιχεία, το θέμα της ψηφιοποίησης των συστημάτων ελέγχου, το θέμα του εγγράφου Α1, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς Γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφύγουμε τις απάτες, να αποφύγουμε τα θέματα του τουρισμού για κοινωνικά θέματα. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε εδώ ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις που κάνει ο κύριος Μπαλάς και πολλές φορές Σήμερα κάποιος πρώτα ψάχνει μια θέση εργασίας μέσω διαδικτύου και κατόπιν αποφασίζει να ε, πάει πάει τόπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ε, διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να μπορέσει ο εργαζόμενος να πάει επιτόπου έτσι ώστε να ψάξει και να βρει τη δουλειά. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι να ενισχυθούν οι προτάσεις του κυρίου Μπαλάς όσον αφορά την ψηφιοποίηση των εγγράφων και τη δημιουργία συνθήκων τέτοιων έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί που ψάχνουν δουλειά να μπορούν να έχουν απαραίτητα στοιχεία και να κάνουν τις πρώτες ε, διεργασίες ε, από τη χώρα διαμονής τους. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά παρόλα αυτά τις προτάσεις του κυρίου Μπελάς για τους ελέγχους. Τα επιδόματα, οι δυνατότητες που προσφέρονται σε κάποιες χώρες σίγουρα προσελκύουν συγκεκριμένους εργαζόμενους σε κάποιες χώρες και όχι σε άλλες. Υπάρχουν σήμερα πολύ συγκεκριμένες ροές, τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσουμε και βλέπουμε σήμερα υποθέσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι οποίες είναι συγκεκριμένες ε, υποθέσεις οι οποίες αφορούν απάτη, καταχρήσεις στα κοινωνικά επιδόματα και στις κοινωνικές παροχές. Θα πρέπει κάθε φορά λοιπόν να ελέγχουμε αν η κάλυψη παραδείγματος χάρη ιατρικών ε, αναγκών, ιατρική περίθελψη, αλλά και τα οικογενειακά επιδόματα και αυτό είναι το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να δείξω. Και ο κύριος Μπαλάς βεβαίως ε, έθεσε κάποιους περιορισμούς όσον αφορά το θέμα της ε, μεταχείρισης των οικογενειακών υποδημάτων, των επιδομάτων παιδιών και κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν ή να μην προσχωρήσουν στην ε, δυνατότητα να βρεθούν κοινά συστήματα για τα οικογενειακά επιδόματα και ιδιαίτερα για τα επιδόματα για τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Η Χέλγα Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία του και βεβαίως με την ψηφιοποίηση έχουμε σήμερα νέες δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα για να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping. Σίγουρα δεν υπάρχει αρκετός διάλογος και θα πρέπει να υπάρχει πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη συνεργασία. Δεν μπορούμε πλέον να δεχόμαστε έγγραφα τα οποία είναι μη γνήσια παραδείγματος χάρη. Επίσης, οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά αργές σήμερα. Στη Φλάνδρα οι εργαζόμενοι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ανταγωνιστικοί, διότι είναι πάρα πολύ ακριβή. Έχουμε δύο χρόνια, μία περίοδο δύο ετών, μέχρι να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους τοπικούς εργαζόμενους. Η εσωτερική αγορά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευτεί και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες που θα επιτρέψουν στους πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα το Brexit. Είμαι πεπισμένη ότι ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλιξης μπορεί να είναι ένας από τους τρόπους να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην, προς την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά συστήματα. Χαίρομαι που η Επιτροπή θέλει να αποφύγει τον ε, τουρισμό, κάτι που είναι μια μάστιγα στον τομέα των κοινωνικών ε, δικαιωμάτων. Τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που δίνεται σαν δώρο μόλις κάποιος περάσει ένα σύνορο χρειάζονται τουλάχιστον τρει μήνες εργασίας στη χώρα φιλοξενίας πριν κάποιος μπορέσει να υποφεληθεί από τα κοινωνικά επιδόματα. Μετά από ένα μήνα δεν μπορεί κανείς να ζητάει κοινωνικά επιδόματα, δεν υπάρχουν καν δεσμοί με τη χώρα στην οποία εργάζεται. Χρειάζεται βεβαίω κωδικοποίηση τη νομολογίας και για τους μη ενεργούς και μη εργαζόμενους και το θέμα των κοινωνικών επιδομάτων που αφορούν την οικογένεια του εργαζόμενου, τα παιδιά του, είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως και τις επιπτώσεις στην ανεργία, το πώς θα ενδυναμώσουμε τους ελέγχους και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για Ευρωπαϊκή Αρχή της Αγοράς Εργασίας και για Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα εργασίας. Είναι πολύ νωρίς για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφευχθούν οι καταχρήσεις, υπάρχουν νέε ευκαιρίες και νομίζω ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και νομίζω ότι θα ακολουθήσει η επικοδομητική συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι στις τροπολογίες 5, 6, 7, 55 και 71 υπάρχουν κάποιες νέες ευκαιρίες που αφορούν τις δυνατότητες που δίνει ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε αυτές οι προτάσεις, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Η τροπολογία 49 θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να δώσει μία λύση σε αυτό που μόλις προανέφερα. Το ερώτημά μου είναι Αυτό ακριβώς δεν προτείνει σήμερα η ευρωπαϊκή πολιτική για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο εισηγητή ε, δεν ε, υποστηρίζει τη δυνατότητα ενός εξαμήνου που μπορεί να επεκταθεί η Επιτροπή θεωρώ εδώ ότι δίνει περισσότερη ευελιξία και είναι πολύ πιο ισορροπημένη η πρότασή της. Επίσης όσον αφορά τη συσσόρευση και όσον αφορά την πρώτη περίοδο, ένας μήνας ή τρεις μήνες, από τη στιγμή που μπορεί κάποιος να απαιτήσει κοινωνικά δικαιώματα. Νομίζω ότι οι τρεις μήνες είναι μια λογική πρόταση Και βεβαίως ο τριμερής διάλογος, η προσπάθεια να βρεθεί ένα ισορροπημένο κείμενο εδώ στην Επιτροπή δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά θα πρέπει κάποιες από τις αναφορές να διαγραφούν, όπως παραδείγματο χάρη η περίοδος των 20 μηνών που υποβάλλεται από μια άλλη τροπολογία. Τροπολογία 13. Το θέμα της δικαιοδοσίας των ε, δικαστηρίων. Καθώς και η τροπολογία 38. Και εδώ θέλουμε να συζητηθούν αυτά τα δύο σημεία. Όσον αφορά τώρα τους ε, μη ενεργά οικονομικούς, ε, εδώ πρέπει να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τον Οργανισμό Εργασίας ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής. Με μεγάλη χαρά θα κοιτάξουμε αυτές τις προτάσεις και δεν προτείνουμε πλήρη διαγραφή. Ε, περίθαλψη για χρόνιες ασθένειες. Στα πλαίσια της ενδοκινοτικής κινητικότητας, Βεβαίως εδώ θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και περίθαλψης και κάποια κράτη-μέλη βεβαίως εδώ το προβλέπουν ήδη. Χρειάζεται εδώ ξεχωριστή, ξεχωριστό κεφάλαιο για το θέμα αυτό. Στην πράξη όσον αφορά τον λεγόμενο κοινωνικό τουρισμό ή τουρισμό για τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά στην πράξη. Θα πρέπει βέβαια να καλύψουμε αδυναμίες που υπάρχουν και νομίζω ότι το κείμενο το κάνει αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξαλείψουμε την λανθασμένη ιδέα ότι υπάρχουν πολλές καταχρήσεις και απάτες που στην πράξη νομίζω δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω πραγματικά να εκφράσω το σεβασμό μου για την εργασία του συναδέλφου, του Γκυγιόν Μπαλάς. Νομίζω ότι και σαν σκιώδη συζυγήτρια της πολιτικής μου ομάδας μπορώ να υποστηρίξω αυτές τις προτάσεις. Νομίζω ότι μας μένει λίγος χρόνος και μπορούμε να επεξεργαστούμε τα σημεία που παραμένουν εκκρεμή. Έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες, αυτές που έχουν σαν σκοπό να στηρίξουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τον συντονισμό τους. Θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος, από όπου και αν προέρχεται και όπου και αν πηγαίνει, να έχει κοινωνική ασφάλιση και να του παρέχεται περίθαλψη να μειώσουμε την ανασφάλεια. Το θέμα των οικογενειακών επιδομάτων, των επιδομάτων τέκνων. Εδώ υπάρχουν προτάσεις για την αναπροσαρμογή αυτών των επιδομάτων. Ο εισηγητής ε, εδώ έχει κάνει κάποιες προτάσεις τις οποίες εμείς στηρίζουμε. το θέμα της ε, ιατρικής περίθαλψης, η πρόταση να υπάρξει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, η πρόταση εδώ είναι τα κράτη-μέλη να υποβάλουν ένα κατάλογο με όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ε, προσφέρουμε, αν θέλετε, επιπλέον ε, δυνατότητες επεξεργασίας του κειμένου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ξεχωριστό κεφάλαιο και νομίζω ότι μπορεί όλα αυτά να ενσωματωθούν στο κεφάλαιο 1 όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά θα πρέπει να ισχύουν βεβαίως οι ίδιες συνθήκες παντού. Θα ήθελα να απευθυνθώ εδώ στον εισηγητή και να του πω ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση γίνεται αναφορά εδώ της οδηγίας και αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Θα δημιουργηθεί νομική ασάφεια. Προτείνω λοιπόν να διαγράψουμε αυτή την αναφορά. Βεβαίως όλοι θέλουμε να περιορίσουμε, να πατάξουμε τις καταχρήσεις και τις απάτες, αλλά έχω την εντύπωση ότι μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να απαντήσουν και να δώσουν τα στοιχεία που ζητούν οι εργαζόμενοι. Η προθεσμία για μένα είναι έξι μήνες. Εδώ υπάρχει μια πρόταση για 24 μήνες και όχι μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για τους εργαζόμενους. Τα επιδόματα τώρα που αφορούν την ανεργία. καθώς το θέμα αυτό για μένα ενσωματώνεται και στην ε, συζήτηση που θα έχουμε για τους μη, ενεργά, μη οικονομικά ε, ενεργούς ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού με τα επιδόματα ανεργίας. Το θέμα είναι πόσο χρονικό διάστημα θέλουμε να προβλέπουμε εδώ για την προηγούμενη εργασία αλλά και για την κάλυψη από τα ταμεία ανεργίας. Η συσσόρευση τώρα των δικαιωμάτων. Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι λαμβάνεται υπόψη από την πρώτη ημέρα της εργασίας ενός εργαζόμενου σε ένα άλλο κράτος μέλος. Θεωρούμε ότι εδώ δεν χρειάζεται κωδικοποίηση για τους ε, μη εργαζόμενους, αλλά ένα από τα σημεία τα οποία εμείς εδώ προτείνουμε είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες να συνεισφέρουν στα ταμεία Κοινωνική ασφάλιση των χωρών στις οποίες διαμένουν και στις οποίες εργάζονται και βεβαίω αυτά τα δικαιώματα να μεταφέρονται όταν αλλάξουν χώρα στην οποία εργάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν ε, τις προθεσμίες και βεβαίως όπως ξέρετε η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους προβλέπει ότι από την πρώτη ημέρα της απόσπασης θα πρέπει να ισχύει η προθεσμία και η περίοδος εργασίας. Πρόκειται για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εμείς εδώ ανησυχούμε λίγο όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση. Η νομολογία Ξέρουμε ότι κάποιες αποφάσεις δεν αναφέρονται στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η νομολογία λοιπόν βεβαίως εξελίσσεται Ποιος είναι οικονομικά μη ενεργός, ο ρυθμός εδώ κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνει διαφορετικά. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ λαμβάνει υπόψη σε κάποιες κατηγορίες όπως τους συνταξιούχους, τους ε, ερευνητές, Κάπω θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε εκ νέου το κείμενο της Επιτροπής που αφορά τους μη ε, ενεργούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι η πρόταση της Επιτροπής μας οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση και ότι δεν προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Το θέμα των επιδομάτων τέκνων, των οικογενειακών επιδομάτων, υπάρχει κάτι που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, είναι το θέμα της εντύπωσης που επικρατεί στην Ευρώπη. Είναι μύθος το ότι υπάρχει εδώ ε, ένας μεγάλος αριθμός καταχρήσεων, και απάτης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, δυσφήμιση, αυτή τη λανθασμένη αντίληψη, γιατί βεβαίως ε, χρειάζονται αποδείξεις, έχουν γίνει πάρα πολλές ε, μελέτες και έρευνες στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την λανθασμένη αντίληψη και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη, και εδώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, να μπει αυτό σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Υπάρχουν και τα επιδόματα αναπηρίας, δεν ξέρω αν θέλω να γίνει ξεχωριστό κεφάλαιο για το θέμα αυτό. Πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας. Τρεις μήνες μας φαίνεται ότι είναι μια πολύ λογική προθεσμία. Το θέμα είναι βεβαίως η καταβολή αυτών των ε, επιδομάτων. Υπάρχουν δυσκολίες. Μάλλον εδώ θα στήριζα την πρόταση της Επιτροπής το θέμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να το κάνουμε. Μιλάτε εδώ και τέσσερα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάποιος από την ομάδα των EFDD. Δυόμιση λεπτά έχετε. Η κυρία Ζωέλ Μελά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα εκπλαγεί ο κύριος Μπαλάς αν του πω ότι δεν συμφωνώ. Όχι επί της αρχής, αλλά μιλάμε για συντονισμό. Υπάρχει ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα, το οποίο δημιουργείται εδώ και δεκαετίας. Η κοινωνική Ευρώπη, η Ευρώπη των εθνών, εδώ και 200 χρόνια δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης από την εποχή του Μπίσμαρκ και υπήρχαν διεθνείς συμβάσεις οι οποίες λειτουργούσαν πολύ ικανοποιητικά με πιστώσεις, με ένα σύστημα εξισορρόπησης και συναλλαγών μεταξύ των συστημάτων αυτών. Υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας. Η κοινωνική Ευρώπη ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, εκρεμεί και σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσει ε, με προσεκτικά βήματα. Αν κοιτάξει κανείς τώρα τους αριθμούς, βλέπει ότι για λιγότερο από 300.000 άτομα μη ενεργά για λιγότερο από 200.000 άνεργους διασυνοριακοί, όπως τη λέμε, εργασία και λιγότερο από 100.000 άτομα τα οποία χρήζουν ιατρικής περίθαλψης σε μια άλλη χώρα. Μιλάμε ιδιαίτερα για χρόνιες ε, ασθένειες. Στη Γαλλία πολλές φορές αυτή η κατηγορία αναλώνει πάνω από το 70% του προϋπολογισμού της, του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν άτομα τα οποία δεν συνεισφέρουν να ε, χρησιμοποιούν ε, ένα τόσο μεγάλο ποσοστό των ποσών και των συστημάτων περίθλαψης. Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται αυστηρότερος έλεγχος. Χρειάζεται ένας έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων. Αυτό μας το επιτρέπει η ψηφιακή τεχνολογία. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί δεν θα πρέπει να πέσουμε σε ένα πάρα πολύ ε, αυστηρό αστυνομικό σύστημα που περιορίζει την ελευθερία των πολιτών. Το δικαίωμα για εργασία δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο και φυσικά θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή, με τον κύριο Μπαλάς ε, και θα του υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας. Η κυρία Μωρά Σαρτιέ, η κυρία Σάντερ, ο κύριος Μαχτά, ο κύριος Λέναρς και εγώ. Η κυρία Ράνκε. Και θα ολοκληρώσουμε τον κατάλογο. Η κυρία Μογά Σαρτιέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τον Γκυγιόν Μπαλάς. Είναι πολύ σημαντική, τεχνική και ουσιαστική η εργασία του για να δημιουργήσουμε την κοινωνική Ευρώπη που εγώ υποστηρίζω. Καταρχήν, η αναθεώρηση αυτού του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι καθαριστικό γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε μια πραγματική προστασία των εργαζομένων. Θα βελτιώσουμε με την έκθεση αυτή την κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών και θα καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Θα επιμείνω εγώ σε τρία σημεία. Πρώτον, Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις επιχειρήσεις που δεν είναι πραγματικά εγκατεστημένες σε μια χώρα. Τις λεγόμενες επιχειρήσεις γραμματοκιβώτιο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνουμε με αυστηρότητα. Και αυτό είναι καθαρά θέμα αξιοπιστίας. Ευχαριστώ πολύ τον συγητή. Δεύτερον, το θέμα της απόσπασης με το έντυπο Α1 της κοινωνικής ασφάλισης και η προθεσμία, πόσοι μήνες δηλαδή, είναι απαραίτητη για να μπορέσει κάποιος να ενσωματωθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής. Θα πρέπει τα δύο κείμενα, το κείμενο του κανονισμού για την κοινωνική ασφάλιση και το κείμενο του κανονισμού για τους αποσπασμένους, να τα επεξεργαστούμε από κοινού. Έχουμε μάλιστα ξεκινήσει αυτή την εργασία με την ε, Ανιέσκα και την κυρία Πρόεδρο. Είναι γνωστή η θέση μου για το θέμα αυτό. Οι έξι μήνες για να ενσωματωθεί κάποιος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πριν την απόσπαση ενός ε, εργαζομένου. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν οι έξι μήνες είναι η σωστή προθεσμία. Θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Τέλος, η τροπολογία 24 για τους δημοσιογράφους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραδείγματο χάρη, δημοσιογράφοι σε μια άλλη χώρα πολλές φορές δεν τους ενσωματώνουμε. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ της έδρας της επιχείρησης και του τόπου στον οποίο πραγματικά εργάζονται. Είναι λοιπόν πολύ καλό που με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε μια λύση σε αυτή την περίπλοκη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Τον Γκυγιώμα Μπαλάς, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική η δουλειά σας. Μακάρι όλοι οι συγγητές να εργαζόταν με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο. Η δουλειά μας θα ήταν ευκολότερη. Μιλήσατε και για την λανθασμένη αντίληψη όσον αφορά τις καταχρήσεις που δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα επιδόματα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να βρούμε τις σωστές λύσεις. Όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας, εγώ συμφωνώ πολύ με τον ε, εισηγητή. Θα πρέπει να δίνονται επιδόματα στην χώρα τις οποίες το σύστημα έχει συνεισφέρει ο εργαζόμενος και ότι τα επιδόματα ανεργίας θα πρέπει να καταβάλλονται για μεγαλύτερη περίοδο και όχι μόνο για τρεις ή έξι μήνες, μέχρι να αλλάξει, αν θέλετε, η κατάσταση και όσο ισχύουν τα κοινωνικά δικαιώματα του εργαζομένου. Και νομίζω ότι εδώ η νομολογία του Δικαστηρίου ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφέστατη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά την συνεισφορά κάποιων εργαζομένων και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός των δικαιωμάτων τους κατ' επέκταση. Η περίοδος που προβλέπεται για την και η αλλαγή που προτείνεται από 24 μήνες σε λιγότερο. Όσον αφορά την συνταξιοδότηση, πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την περίοδο των 24 μηνών. Αυτή είναι η απόψή μου. Είμαι κατά της πρότασης να υπάρχουν έξι μήνες το σύστημα της χώρας υποδοχής πριν ξεκινήσει η απόσπαση. Αυτή η πρόταση πραγματικά με βρίσκει αντίθετη. Θεωρώ ότι είναι ένα εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία. η ανεξάρτητη εργαζομένοι δεν μπορούν να αντικαθιστούν τους υπαλλήλους. Αυτό είναι μια παράλογη πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία του Γκυγιον Μπάλλας και να τον ευχαριστήσω διότι ενσωμάτωσε κάποια σημεία τα οποία κατά την άποψή μας είναι σημαντικά. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Η κατάσταση, και επέμενε ο Γκεγιόμ, η κατάσταση των εργαζομένων των διασυνοριακών. Βεβαίως, εάν είναι λογικό και κατανοητό ότι το κράτο μέλος το οποίο ε, έχει εισπράξει τα χρήματα της κοινωνικής ασφάλισης να πρέπει και να τα καταβάλει, είναι σημαντικό και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στους διασυνοριακούς εργαζόμενους που έχουν ε, ως χαρακτηριστικό την κινητικότητα και φτιάχνουν την καθημερινή Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο διότι στις περιοχές που βρίσκονται φτιάχνουν την Ευρώπη περισσότερο από άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να, λάβουμε, να βρούμε μία λύση για αυτούς λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις και να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο ώστε οι δυσενεργειακοί εργαζόμενοι να μπορέσουν να εξαρτηθούν από μια δημόσια αρχή απασχόλησης ε, η οποία θα είναι κοντά στον τόπο στον οποίο εργάζονται. Στην περιοχή μου, στην Γαλλία, ξέρουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται στη Γερμανία. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτή η υπηρεσία που θα χειρίζεται όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι δύσκολα. Κάποιοι που να μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην οποία εργάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι και να γνωρίζουν τα συστήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν σε διασυνοριακό επίπεδο κάποιου τέτοιου υπηρεσίες. Στην περιοχή μου υπάρχουν ε, πάρα πολλοί, αν θέλετε, ε, ο ΑΕΔ, τέτοιου είδους υπηρεσίες, γαλλογερμανικές. Με κάποιο τρόπο λοιπόν θα πρέπει να το διευθετήσουμε αυτό το θέμα ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίκτυο ΕΡΕΣ όπως λέγεται στα αλληλικά. Ακόμη κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε για την ε, ψηφιοποίηση. Με ενθουσιάζουν όλες αυτές οι προτάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με την ψηφιοποίηση αλλά να προσέξουμε να μην δημιουργηθούν ε, επικαλύψεις, διότι προτείνονται διάφορες ε, ε, οργανισμοί, διάφοροι φορείς και διάφορα συστήματα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά, αλλά ίσως έχουμε επικαλύψεις. Ο κύριος Μαρτά, πολύ σύντομα. Δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Μπάλας για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους και εγώ. Και βεβαίως με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Μένω στην ε, Σαββοία, δίπλα στην Ελβετία. Πολλοί ε, Γάλλοι λοιπόν πηγαίνουν να εργαστούν στην Ελβετία. Τώρα, το επίδομα ανεργίας, το κατόφλι αυτό των 12 μηνών. Μετά από τους 12 ε, μήνες λέτε ότι η χώρα υποδοχής θα πρέπει να το καταβάλει. Τι γίνεται όμως με την περίπτωση της Ελβετίας, η οποία είναι, ε, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι Σέγγεν. Δεύτερη ερώτηση, στην οποία θέλω απάντηση. Αυτό το κατόφλι των 12 μηνών είναι ευαίσθητος αριθμός. Εάν ε, αναφερθούμε στο ΡΟΜ 1, δεν θα έπρεπε να δούμε, δεν θα έπρεπε να δώσουμε την επιλογή στον εργαζόμενο να διαλέξει το επίδομα ανεργίας στη χώρα που είναι πιο θετική για αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία που επιτέλεσε για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η πραγματική πρόκληση αυτού του κανονισμού είναι η εξή. Θέλουμε να αποφευθεί οποιαδήποτε κατάχρηση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι όμως πολύ σημαντικό να είμαστε και δίκαιοι για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, ώστε να έχουν, δώσουμε όλες τις ε, δυνατότητες ε, να επωφεληθούν από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης χώρας στην οποία εργάζονται, χωρίς να δημιουργήσουμε εμπόδια. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, οι 12 μήνες, η προθεσμία αυτή την οποία προβλέπει η Επιτροπή. Ενδιαφέρον είναι αυτό που λέγεται, αλλά είναι ίσως και κάπως ε, αφαίρετο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται 20 χρόνια στην Ολλανδία, πηγαίνουν ένα χρόνο στη Γερμανία και με θα μπορούσαν να ζητήσουν ε, να επωφεληθούν ε, των παροχών της γερμανικής κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Επίσης, συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν για τις διασυνοριακές περιοχές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυθαίρετα να επιλέξουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να σκεφτούμε το όλο θέμα των εργαζομένων και πώς θα συνεργαστούν τα κράτη-μέλη για να διευθετήσουν τέτοιου είδους θέματα. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δήλωσης όλων αυτών των θεμάτων μιας χώρας προς την άλλη. Πώς θα κάνουμε τον υπολογισμό των πριν ή των επιδομάτων που πρέπει να καταβάλλονται. Στη δική μου την περιοχή υπάρχουν τέτοιου είδου ερωτηματικά. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης Οι Γερμανοί επιτρέπουν την εργασία μόνο για 15 ώρε εβδομαδιαίως για να παίρνουν κάποια κοινωνικά επιδόματα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, είναι τόσο διαφορετικά τα συστήματα. Επίσης, τι γίνεται σε επίπεδο κάθε χώρας με τα συστήματα διαφορετικά κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συντονιστούμε. Όσον αφορά τις αναπροσαρμογές των οικογενειακών επιδομάτων και τα επιδόματα που δίνουμε στους ε, οικονομικά ανενεργούς. Διαφωνώ με τον ε, ε, εισηγητή, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να πω κάτι σε σχέση με ένα θέμα που αφορά που αφορά το τι γίνεται με τα επιδόματα για τα παιδιά και πώς γίνεται η προσαρμογή αυτών των επιδομάτων. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αν το παιδί ζει σε μια χώρα με χαμηλό κόστος διαβίωσης, τότε είναι κάτι διαφορετικό από ότι αν ζούσε σε μια χώρα που έχει υψηλότερο κόστος διαβίωσης. Αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη οι εξοικονομήσεις του, του κόστους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεράστιο διοικητικό άχθος. Και είναι μια πολιτική που υπονομεύει την αξιοπιστία, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μην υποχωρήσουμε έναντι του λαϊκισμού και θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ δίνω 1,5 λεπτό στον εαυτό μου, λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο για την χρόνια περίθαλψη, θα πρέπει να καθορίσουμε επακριβώς τι καλύπτει, ποιος ακριβώς είναι ο ορισμός. Αυτή είναι η αφετηρία. Και το πιο κρίσιμο θέμα είναι η προστασία και η, ε, ε, η βοήθεια για τους ηλικιωμένους και η περίθευση τους ηλικιωμένους ε, και κατά πόσο είναι εξαγώγημες αυτές οι υπηρεσίες. Όλη αυτή η υποστήριξη που αφορά προσωπική βοήθεια και περίθαλψη ηλικιωμένων δεν είναι κάτι που μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη χώρα χωρίς αύξηση των δαπανών ε, για το κράτος. Και δεν θα πρέπει να μην κυριαρχήσει αυτό το θέμα στη συζήτηση. Να υπογραμμίσω επίσης ότι είναι σημαντική η προσέγγιση του κυρίου Μπάρα αφορά τον περίπλοκο χαρακτήρα της δικαιοδοσίας, το κοινωνικό dumping κλπ. και τους ε, μη δραστηριοποιημένους οικονομικά πολίτες. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τον κατάλογο και ο κ. Κορέ λοιπόν θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Σάντζεφ, θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, διότι είναι σημαντικά τα θέματα. Στις ε, τροπολογίες θα συμπεριληφθούν πολλές αλλαγές και νομίζω ότι δύο λεπτά ο καθένας δεν μας επέτρεψε να πούμε ό,τι θέλαμε να πούμε. Ας οργανωθούμε λοιπόν παρακαλώ για να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Πολύ καλή η πρότασή σας. Νομίζω ότι θα το ξαναθέσουμε το θέμα υποσυζήτηση, διότι πραγματικά νομίζω ότι είναι πρωταρχική σημασία να το συζητήσουμε και ε, γιατί είναι σημαντικό και μακροπρόθεσμα και για μας για τις επόμενες ευρωπαϊκές ε, ε, εκλογές. Θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουρέλ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπάλλας, καθώς και όλους τους παρεμβαίνοντες. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να πω ότι αυτό το οποίο είναι ενθαρρυντικό στο φάκελο αυτό είναι από τότε που ανέλαβε ως εισηγητής ο κύριος Μπάλας με διάφορες ακρεάσεις που είχατε. Εδώ είδαμε ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συνένεση όσον αφορά την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλη συνένεση δεν σημαίνει πλήρης ε, ε, συμφωνία. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες και από τον Ισογητή και από άλλες πολιτικές ομάδες. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά σύντομα. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που οποίο ήδη γνωρίζετε. Ίσως προχωρά ανακεφάλαιο και το Συμβούλιο. Πρόσφατα πρέπει να πω ότι για δύο κεφάλαια υιοθέτησε μια κοινή προσέγγιση και προβλέπεται στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο να επιτευχθεί ακόμη περαιτέρω συμφωνία και κοινή προσέγγιση και σε κάποια άλλα κεφάλαια. Λαμβάνοντας υπόψη και το δικό σας ε, τα δικά σας χρονοδιαγράμματα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να αρχίσει ο τριμερής διάλογος στις αρχές του επομένου εξαμήνου. Και όπως υπογράμμισαν όλοι οι παρεμβαίνοντες, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι θέλουμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα των εργαζομένων χωρίς να χάνουν τα δικαιώματα των οποίων χαίρουν όταν πάνε σε άλλη χώρα να εργαστούν. Και θα πρέπει να δοθούν όλα τα μέσα στις δημόσιες διοικήσεις για να καταπολεμούσουν απάτη και κατάχρηση από κάποιους. Ε, χαιρετίζει λοιπόν η Επιτροπή το γεγονός ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στην επεξεργασία αυτής της πρότασης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε λοιπόν με νέο χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε ότι μία ακόμη συνεδρίαση δεν θα οδηγήσει σε αλλαγέ στο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί για την ε, προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών, αλλά εν πάση περιπτώσει το συντομότερο δυνατό όταν ε, βρούμε χρόνο θα προχωρήσουμε ώστε όλοι όσοι δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο σήμερα να μπορέσουν να το κάνουν. Κύριε Μπάλας. Ποια είναι η δική σας θέση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν στην ε, συζήτηση. Κύριε Λούντεφτσα, και εγώ υποστηρίζω την απόψή σας. Αν πραγματικά μπορέσουμε να οργανώσουμε και μια νέα συνεδρίαση, χαίρομαι ιδιαίτερους. Διαφορετικά. Εγώ θα είμαι ε, διαθέσιμος και πέραν του χρόνου που μπορώ να με όλους τους και τους όχι με τον καθένα χωριστά, δεν έχω τόσο χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων, χωρίς βεβαίως να μην δώσω προτεραιότητα στους κοινωνικούς εισηγητές, πράγμα το οποίο είναι σύνηθες και λογικό. Ο κύριος Κουρέλ από την Επιτροπή κυρίστηκε σωστά το θέμα. Είπε ότι όντως εκφράστηκαν διάφορες απόψεις για διάφορες αποκλίνουσες νόμες και είδαμε ότι τελικά το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι να έχουμε συγκλίνουσες απόψεις σε πολλά θέματα. Παρά το γεγονός ότι θα προσπαθήσει, κύριε Κουρέλ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του την πρόταση αυτή και να παρουσιάσει μια ενιαία θέση στα πλαίσια του δυνατού. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις αρχίζοντας με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Αρχή. Ναι, σε ένα νομοθετικό κείμενο μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Θα ήθελα παρόλα αυτά να προσθέσω ότι κάθε φορά που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγγέλει κάτι το πολύ σημαντικό και είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κοινωνικών Θεμάτων να μπορεί να εκφράσει την απόψή τη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό. Γι' αυτό ας μην αφήσουμε κατά... Μην, ε, ε, ας αφήσουμε κατά μέρος κάποιες ε, έννοιες, κάποιες λέξεις πίσω από τις οποίες δεν κρύβεται σχεδόν τίποτε το θετικό. Διότι δεν συνάδουν αυτά με την καλή κοινωνική ε, θέση που θέλουμε να δώσουμε στην Ευρώπη. Για τις ερωτήσεις που κάνατε τώρα για την Ελβετία. Για το IMF. Δεν το Ρώμα, δεν το γνωρίζω αυτό που είπατε, θα το εξετάσω. Σίγουρα υπάρχουν όμως ένα διαφυγόν κέρδο για κάποιους, θα το εξετάσουμε Δηλαδή ξέρουμε ότι στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν ε, ε, ένα διαφικό κέλος 600 ε, εκατομμυρίων. Την αφορά αυτό το θέμα την Ελβετία, την Ευρωπαϊκή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως το Λίχτενστάιν, όσον αφορά τους διασυνοριακούς εργάτους. Κύριε Σάντερς, πού είναι Πού είναι η κυρία Σάντερς. Όντως θα πρέπει να εξετάσουμε το EURES. Αν μπορεί δηλαδή το EURES, το RES να συνεργαστεί μαζί μας και να δημιουργήσουν κάποια ε, θετικό θέμα για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους να είναι να συνεισφέρει θετικά και να συμμετάσχει στο όλο θέμα. Ε, εξαιρετική ιδέα, εξαιρετική δεν την είχα σκεφτεί και θα την μελετήσω περαιτέρω. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά το σύνολο της πρότασης, ή της πρότασης της Επιτροπής ή της πρότασης που υπέβαλα εγώ. Κάποιοι υποστηρίζουν λοιπόν τις δικές μου προτάσεις, όπως Φερρυπίν στο θέμα της εξαγωγής των ε, δικαιωμάτων σε ε, επιδόματα ανεργίας άλλοι για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Άλλοι είναι εντελώς αντίθετοι. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν αντιθέτεις που ξεπερνούν και τα πολιτικά, ε, τις πολιτικές ομάδες και εξαρτώνται ίσως ε, από την κάθε εθνική νομοθεσία και κάθε εθνικό σύστημα. Θα πρέπει να βρούμε μία μέση οδό. Εάν μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν κυρίως στο θέμα της ψηφιοποίησης, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η κυρία Άρκιν είπε ποια είναι η απόψή της, είπε δεν θα πρέπει να προσθέσουμε πολλά πράγματα και νέους φορείς, υπάρχει το SSE το οποίο κάποια στιγμή θα τεθεί σε εφαρμογή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι σήμερα δεν ξέρουμε τι είναι το SSE. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο μια πλατφόρμα δεδομένων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα και γι' αυτό το λόγο πήρα το παράδειγμα του βελγικού συστήματος να έχουμε σε μία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων που διαθέσουμε, ώστε οι διοικητικές αρχές να είναι πλήρως ενημερωμένες. Διαφορετικά, ως συνήθως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μία πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί αλλά θα υποχρησιμοποιείται. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε το SSE, αλλά να το ενισχύσουμε και να του προσδώσουμε πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των διαφορετικών κεφαλαίων για, ε, μακροχρόν, για τη μακροχρόνια υγειονομική κάλυψη και ιατρική περίθαλψη. Όταν εδώ στο ε, hearing που είχαμε κάνει στην ακρόαση των ε, Ευρωπαϊκής ε, Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ήθελε να υπάρχουν όλα αυτά σε διαφορετικό κεφάλαιο. Εγώ εμπνεύστηκα πάρα πολύ. Να ζητήσουμε όμως να συνεργαστεί μαζί μας για το θέμα αυτό. Θα πρέπει επίση και η κοινωνική εταίροι. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε διαφορετικό κεφάλαιο, αλλά είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση για τα θέματα αυτά. Τελειώνω τώρα με θέματα τα οποία αφορούν την αναπροσαρμογή και την κωδικοποίηση. Και θα πω και δύο λόγια για κάποιο άλλο θέμα. Το θέμα της κωδικοποίησης. Δεν είναι υπέρ το Συμβούλιο σήμερα. Το διαπιστώνουμε αυτό. Μπορούμε να το κατανοήσουμε και τα επιχειρήματα που προβάλλονται για την κωδικοποίηση, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, να γνωρίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Εγώ, και βεβαίως είμαι ανοιχτός για οποιαδήποτε συζήτηση, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μία μερική κωδικοποίηση, Ας αφήσουμε στο νομοθέτη να ασκήσει τα καθήκοντά του, αλλά είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συζήτηση. Τώρα, το θέμα τη προσαρμογή. Δεν μίλησα και δεν θα έπρεπε να μιλήσω, διότι δεν υπάρχει επί αυτού του θέματος καμία πρόταση εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες, κάποιες χώρες που σήμερα θα ήθελαν να γίνει αυτή η προσαρμογή. Όταν συζητούμε όμως με αυτές τις χώρες, διαπιστώνουμε ότι είναι για να πληρώνουν λιγότερα. Αυτό όμως έχει και άλλα αποτελέσματα. Φερρυπίν, έχουμε αλλοδαπούς ε, γονείς που εργάζονται σε μία χώρα και θέλουν να έρθουν τα παιδιά τους να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά τι θα τους κοστίσει. Και σήμερα όντως η αναπροσαρμογή θα είναι γραφειοκρατική, αναποτελεσματική και πολύ δαπανηρή. Δεν θέλω λοιπόν να πάω πιο μακριά από αυτά τα οποία πρότεινε επί του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος πάντων, δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Θα μελετήσω όλα όσα ελέγχθησαν. Θα συναντηθώ με τον καθένα από τους χειώδεις ηγητές και θα γίνει η συζήτηση η συνολική που θα γίνει τον Ιανουάριο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα διεξοδικά ως ομάδα. Γι' αυτό θα ζητήσουμε στην γραμματεία να προσπαθήσει να μας βρει μια κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Διότι, το συντομότερο δυνατό αυτό, διότι γνωρίζουμε τα προβλήματα και θα πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές. Οι προθεσμίες όμως δεν αλλάζουν, έτσι όπως τις είχαμε ορίσει, δηλαδή 10 Ιανουαρίου προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, 21 με 22 Φεβρουαρίου εξέταση των τροπολογιών, έγκριση στις 19 Ιουνίου στην ε, ε, Επιτροπή μας. Αυτά προς το παρόν και τώρα προχωράμε με το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρολά, τον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω, αλλά θα το κάνω, να υπενθυμίσω ότι πρώτη λόγος της ημότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος που έχει σχέση με το επάγγελμα του καθενός. Κάθε ώρα, κάθε μέρα μισθωτοί πεθαίνουν εξαιτίας της Έκθεσή τους στην εργασία σε κίνδυνο. Θα ήθελα να πω ότι χρειάστηκε στην Επιτροπή 10 χρόνια που ξανά το φάκελο αυτό για να βελτιώσει τη σχετική οδηγία. Ο στόχος της κυρίας Τέσεν, της Επιτρόπου, είναι να κάνει τρεις αναθεωρητικές προτάσεις ώστε να μπορέσουν να αναπροσαρμοστούν οι εκθέσεις σε καρκινογόνες και ε, ουσίες βάσει των επιστημονικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, να μπούμε σε έναν μηχανισμό διαρκούς αναπροσαρμογής συγγνώμη, των διαφορών ανωτάτων πεδίων. Πιστεύω ότι αυτό θέλει και η Επιτροπή και ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος. Τώρα, η, η πρόεδρος ήταν και η συγγήτριά μας για το θέμα αυτό. Με αυστηρότητα, πραγματισμό και φιλοδοξία θα πρέπει να προχωρήσουμε, διότι θα πρέπει να βασιστούμε με, στα απορίσματα στα οποία καταλήγουν οι επιστημονικές περιοχές. Η φιλοδοξία μας θα είναι να προστατεύσουμε την υγεία όλων των εργαζομένων και με πραγματισμό λαμβάνοντας υπόψη τι συμβαίνει στις διάφορες επιχειρήσεις που έχουν τα οικονομικά του συμφέροντα και έχουν και τις τεχνολογικές εκκλήσεις. Και βεβαίως όλα αυτά με τη συνένεση των κοινωνικών εταίρων. Χαιρετίζω την Επιτροπή διότι έκανε σωστά τη δουλειά της πριν να μας υποβάλει προτάσεις και συστάσεις ε, μετά από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν συμβουλευτικές και επιστημονικές και τεχνικού περιεχομέ... τεχνικής φύσεως επιτροπές για να καταλήξουμε σε διάφορα κατόφλια. Και υποστηρίζω πολλές από τις προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή, αλλά θα καταθέσω διάφορες προπολογίε για να προστατεύσουμε καλύτερα τους ε, εργαζόμενους που εκτίθενται στα διάφορα καυσαέρια των κινητήρων δίζελ και στο πολυκυκλικούς αρωματικούς αδρογονανθάκων. Ζητώ συγγνώμη από τους διεθμινείς. Θα τους, ονομα... θα τους ε, λέγω με, το... με τη στιμογραφία τους. Πάει στα ελληνικά. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τα ανώτατα κατόφλια έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει το συντομότερο εργαστό να επεξεργάζεται το όλο θέμα αυτό η Επιτροπή και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητώ στο σχέδιο έκθεσής μου. Επίσης θα ήθελα να ασχοληθούμε με όλου των ειδών τα καυσαέρια και να μην περιοριστούμε μόνο στο βενζοπυρένιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προβλέπει και στις γενικές καθεδρίες γραμμές του το Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα τα καυσαέρια των γεννητήσεων «Δίζελ» οι προσδοκίες παραμένουν μεγάλες εκ μέρους των εργαζομένων. Στην ετελειακή της έκθεση η Επιτροπή δεν προτείνει να συμπεριληφθούν στην επόμενη αναθεώρηση τα καυσαέρια κινητήζων δίζελ. Λυπούμε, διότι 3,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στα καυσαέρια των κινητήρων δίζελ. Και περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άτομα πραγματικά ε, πεθαίνουν, διότι εκτίθενται σε τέτοιου είδους δηλητηριώδη ε, καυσαέρια. Γι' αυτό θα ήθελα τα καυσαέρια, οι φομπές καυσαερίων κινητήρων diesel να συμπεριληφθούν με 50 ε, μικρογραμμάρια ανά ε, κυβικό μέτρο. Ανώτατο όριο πράγμα το οποίο ξεπερνάει και τους μέσους όρους συνήθως. Επίσης, τελειώνοντας, θα ήθελα να επιμείνω σε δύο άλλα στοιχεία. Η πρόληψη και η έλεγχη. Σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η πιο σημαντική λέξη είναι η πρόληψη, που σημαίνει ότι πρέπει να σεβόμαστε πάρα πολλούς κανόνες και να κάνουμε σωστούς ελέγχους. Οι διάφορες τομεακές συμφωνίες που έχουν κάνει με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν να επιτρέψουν εργοδότες στους εργαζόμενους να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι η επικινδυνότητα των διαφόρων ε, ε, ουσιών και υλικών τα οποία χειρίζονται για να είναι προσεκτικοί. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη στις συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο για τους εργαζομένους. Και θα ήθελα να συμπεριλάβω σε όλα αυτά τα οποία λέω στα πλαίσια της συμφωνίας νέψη και το κρυσταλλικό πυρίτιο το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Τώρα, στις διάφορες επιχειρήσεις οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προορατικά θα πρέπει να δουν πώς θα μπορέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προστατεύσουν την υγεία των εργαζομένων. Και έτσι όλοι κερδίζουμε, διότι προστατεύονται οι εργαζόμενοι, λειτουργούν περισσότερα, ε, καλύτερα οι επιχειρήσεις και ο νομοθέτης μπορεί πιο εύκολα να κάνει τις κατάλληλες και πιο ρεαλιστικές προτάσεις. Η αναθεώρηση βεβαίω τη ε, οδηγία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και του ελέγχου που πρέπει να γίνονται στι διάφορε επιχειρήσει από τι υπεύθυνε αρχέ. Οι έλεγχοι αυτοί δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στην επιβολή κυρώσεων από τι επιχειρήσει που δεν σέβονται τι ε, σχετικέ διατάξει. Θα πρέπει να εντοπίζουν τι αιτίε του μη σεβασμού της οδηγίας και να κάνουν προτάσεις για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα μια τέτοιου είδους οδηγίας, κυρίως στις ΜΜΕ. Για μένα ο έλεγχος, ναι, μπορεί να έχει και κυρωτικό χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει κυρίως να έχει ως πρώτο στόχο την ευαισθητοποίηση και συνοδευτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη περισσότερο και καλύτερα την υγεία των εργαζομένων. Αυτά έχω να πω. Όπως κάναμε και την πρώτη φορά, πιστεύω ότι επιτύχαμε μέχρι τώρα σε αυτά τα οποία κάναμε από κοινού. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε από κοινού ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις στο πρόβλημα αυτό που είναι τόσο σημαντικό για τι επιχειρήσεις και του εργαζόμενου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρολά. Θα μιλήσω στη θέση σκιωδών των σκιωδών και θα επιβεβαιώσω αυτά που είπατε. Καταρχάς ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Πάρα πολύ καλή έκθεση. Μάθαμε πολλά κατά τη διάρκεια της πρώτης της οδηγίας. Μάθαμε πολλά για τις ουσίες και για το πού πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες της Επιτροπής για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Συμφωνώ απολύτως με την πρόταση του κ. Ρολάν. Η συμπερίληψη του ντίζελ είναι ύψης της σημασίας. Συμφωνώ με την επιλογή του που χρησιμοποιεί τον άνθρακα, τον βασικό άνθρακα για την εξάτμιση από κινητήρα diesel. Καλή επιλογή. Καλύπτει κάθε μορφή diesel και τις παλιές μορφές που είναι οι πιο επικίνδυνες. Και αυτή είναι και σύσταση της ε, Επιτροπής ΣΚΟΛ βάσης, βάσει των συστάσεων σε λόγω επιτροπής να συζητήσουμε και οριακές τιμές για ε, το αζωτούχα, ε, οξύδια, το αζωτούχα οξύδια για να μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλες μορφές ρήπανσης από κινητήρες δίζελ. Αυτή η άποψη βασίζεται επί της νομοτήσεως σκολ για τους κινητήρες δίζελ. Δεν δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ αυτή τη γνωμοδότηση. Παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Όλες οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής αυτής της ΚΟΑΛ πρέπει να δημοσιευτούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Ακόμα και αυτές που είχαν συνταχθεί επί της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόσο. Είναι προς το συμφέρον του κοινού που πληρώνει και είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε σε αυτή την της οδηγίας, όμως πρέπει να τεθεί το ζήτημα. Αφορά το μέλλον των εργασιών ε, της Επιτροπής ΚΟΛ. Δεν έχουν αναλάβει κάποια καινούργια εργασία και θα αναδιοργανωθεί η Επιτροπή. Ε, είναι πολύ σημαντικό το έργο της Επιτροπής ΣΚΟΛ και για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο. Και αν αναδιοργανωθεί, δεν θα πρέπει να χάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη της. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε τις οριακές τιμές, Φερρυπίν, χωρίς επιδημιολόγους και τούτου λεχθέντος υποστηρίζουμε ένθερμα την πρόταση του κυρίου Ρόλαμ και τη συμπερίληψη των κινητήρων δίζελ. Η ε, κυρία Μάκινταρ είναι η επόμενη θα πάρει το λόγο, ο σκιώδης εισηγήτρια. Α, δεν είναι εδώ. Η ε, κυρία Στίβενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Μάκινταρ που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Καταρχάς, καλωσορίζω τη δεύτερη φάση των τροπολογιών. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο εκθέσεώς του. Οι οριακέ τιμέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποτελέσματα πολλών ετών λεπτομερών εργασιών και αξιολογήσεων και δοκιμών. Υπάρχει αυστηρή διαδικασία για τον καθορισμό των τιμών. Βασίζονται σε στοιχεία, είναι αναλογικά προ μετρήσιμα όρια και μπορούμε να τα πετύχουμε. Πιστεύω ότι η δραστηριοποίηση για τη μείωση του αριθμού των θανάτων σε περιπτώσεις εκθέσεως σε καρκινογόνες ουσίες που βλάπτουν την υγεία και εκθέσω άλλε επικίνδυνε ουσίε είναι υψή τη σημασία. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε στον έλεγχο επαγγελ... της επαγγελματικής εκθέσεως στις κακινογόνε ουσίες. Αυτό οδηγεί σε αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων. Πρέπει να τονίσουμε την εφαρμογή ορθών πρακτικών ελέγχου. Επίση πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το ρόλο των καλών πρακτικών όπως είναι οι πρακτικές του NEPSI, του κοινωνικού, της Συμφωνίας του Κοινωνικού Διαλόγου και να υποστηρίξουμε την εφαρμογή της οδηγίας για τα καρκινογόνα και τα ε, μεταλλαξιογόνα. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι όλες οι εκθέσεις της ουσίας ε, ελέγχονται και η έκθεση είναι στο χαμηλότερο δυνατό όριο. Οι ηρικές τιμές θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο που ελέγχουν τους κινδύνους έκθεσης επιβλαβής ουσίας. Τελικός στόχος τα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Χαμηλότερα από τα επίπεδα που καθορίζει η νομοθεσία, παραδείγματο χάρη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ενεργώ να επενδύσουν στην επιστήμη, να ενθαρρύνουν τι επιχειρήσει και τι εταιρείε συνεχώ να προσπαθούν για τα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα έκθεση. Δεν μπορούμε αυθαίρετα να καθορίζουμε επίπεδα που είναι τόσο χαμηλά που δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε. Η οδήποτε νέα πρόταση για αλλαγή των οριακών τιμών θα πρέπει να υπόκειται στην ίδια αυστηρή αξιολόγηση όπως και τον καθορισμό των τιμών. Παρομοίω, η αδίποτε πρόταση για πρόσθεση ουσιών θα πρέπει να υπόκειται στην ίδια διαδικασία. Γι' αυτό το σκοπό η ομάδα μου έχει κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την πρόταση συγγητού να οι οριακές τιμές να καθοριστούν για έκθεση επαγγελματική στις εκπομπές από κινητήρες ε, diesel. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας αυτή την πρόταση, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει αυτέ τι οριακέ τιμέ για κάποιου πρακτικού και νομικού λόγου, όπω καθορίζεται στο τμήμα 4, 2, 3 ε, της αξιολογήσεως αντιχτύπου που συνοδεύει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν αυτού, η, ΕΣΥ, η ΣΕΟΛ ε, έχει συμπεράνει ότι θα πρέπει να καθοριστούν όρια για την έκθεση των εργαζομένων σε, αυτά, σε αυτές τις ουσίες, αλλά είναι κάτι ανέφικτο για την ώρα. Μπορούμε να βρούμε όσο κάποια λύση τελικά Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε τη συμπε... τον δεχόμενο συμπερίληψη θέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τι εργασίε για να καλυφθούν οι ανησυχίε που έχουν εκφραστεί και να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υποβληθεί μια νέα πρόταση για οριακές τιμέ. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μελετηθεί κατά πόσο είναι να εφαρμοστούν τα μέτρα που πρέπει να είναι ανάλογα για να πετύχουμε αποτελέσματα ε, ε, πραγματικά ευχαριστούμε τον εισηγητή για το έργο του και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες που θα αντικατοπτρίζουν τη θέση της ε, ομάδας μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαμπόμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά, διότι έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω τον κύριο Λάου ε, προσωπικά πρόσωπο με πρόσωπο. Ως της ομάδας για το θέμα αυτό, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο για την εργασία που επιτέλεσε. Και πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνάδελφος στην πρώτη του πρόταση έκαναν πολύ καλή με την πρότασή του ο συνάδελφος κύριος Μωρά έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση του συστήματος. Βεβαίω, συμφωνώ με την πρωτοβουλία που έλαβε η Επιτροπή και με το πνεύμα και με το στόχο που θέλει να πραγματοποιήσει. Είμαι λοιπόν σύμφωνοι με την ε, πρόταση που έκανε και ο κύριος Ρολά και θέλουμε να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως απομακρυνόμαστε από ένα θέμα ηθικής. Δηλαδή, αν ε, δεν προχωρήσουμε προς μία κατεύθυνση, θα μας πει κάποιος ότι ε, αναπτύσσουμε αντιεργατικό πνεύμα. Και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει παρόλα αυτά ότι το πρώτο μας μέλημα είναι να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ τεχνικό το θέμα, να προχωρήσουμε με πνεύμα εξισορρόπησης όλων των στοιχείων. Βεβαίως υπάρχουν οι τεχνικές εξελίξεις, τις οποίες γνωρίζουμε, Και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι βελτιώνονται τα πράγματα παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν πολλά προβλήματα. Αυτό το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στο να βελτιώσουμε τα ανώτατα όρια είναι να μπορούμε να κάνουμε πραγματικές μετρήσεις. Δηλαδή, οι τεχνολογικές εξελίξεις μας βοηθούν να μετρήσουμε σωστά τα ανώτατα όρια για να τα καθορίσουμε. Τώρα, στο πλαίσιο του ότι θα πρέπει να βελτιώνουμε πάντα τα πράγματα, να βελτιώνουμε την ορθολογική χρήση της αρχής προφύλαξης και προστασίας και να μην μπαίνουμε σε θεωρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία γίνονται στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου δεδομένου ότι αυτοί στους οποίους ενδιαφέρει η υγεία των εργαζομένων είναι και οι εργαζόμενοι και κυρίως στα πλαίσια των ΜΜΕ οι ε, επιχειρηματίες, οι διευθυντές των επιχειρήσεων, οι οποίοι κυρίως επαναλαμβάνουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ίδιοι είναι εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι και εργαζόμενοι. Το να φτάσουμε λοιπόν σε βέλτιστα αποτελέσματα στα πλαίσια του κοινωνικού ε, διαλόγου είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Θα πρέπει όμως να δούμε κάποια συγκεκριμένα θέματα όπως ανέφερε και ο συνάδελφος. Το θέμα των ε, εκπομπών καυσαερίων από τους κινητήρες diesel και σε άλλα θέματα. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτά με γνώση του θέματος και με επικοδομητικό τρόπο. Και βεβαίως θα το κάνουμε αυτό αφού έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση με τους συναδέλφους, με τους επιχειρηματίες, με τα συνδικάτα. Όσον αφορά τα θέματα αυτά των καυσαερίων, των ζωντήρων, θα πρέπει να μας πει πιο, με πιο λεπτομεριακό και εμπεριστατωμένο τρόπο η Κομισιό τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε διασταυρώσει τα στοιχεία, τα απαραίτητα, τα οποία πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ανάλογα με τους κινητήρες αυτούς που είναι και πολύ διαφορετικοί ανάλογα με την ε, ε, σημασία τους για να προχωρήσουμε με τρόπο σωστό και δίκαιο. Ευχαριστώ. Συνεχίζει ο κ. Λεγιάχικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω μετά όσα είπε ο κ. Ρολόν. Χαιρετίζω και το έργο του. Διορθώνει σημαντικότατο κενό. Είναι τη συμπερίληψη στην αναθεώρηση της οδηγίας του ντίζελ και των συνεπειών αυτού. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την υγεία 19 εκατομμυρίων εργαζομένων, οδηγών, εκείνων που ασχολούνται με την παράδοση εμπορευμάτων που εκτίθενται πολύ συχνά δύο επιχειρήματα προβάλλονται για να αποκλειστούν οι εκπομπές ε, diesel από την αναθεώρηση. Πρώτο επιχείρημα. Οι νέοι κινητήρες πλέον είναι πιο αποδοτικοί και ρηπαίνουν λιγότερο. Δυστυχώς η εμπειρία καταδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερες ε, αμφιβολίες από αυτό που επιτρέπεται Δεύτερον επιχείρημα, ότι το βενζοπυρένιο, μια μία από τις ουσίες, είναι ε, απειροελάχιστη ε, ουσία από, τα, από τους αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και μελετήθηκαν ελάχιστα αυτές οι ουσίες από πλευράς τοξικολογικής. Στην πρόταση αναθεωρήσεως εξάλλου η έκθεση σε αυτούς τους υδρογονάνθρακες, τους πολυκυκλούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, δεν περιορίζεται παρά μόνο στην ε, έκθεση του δέρματος στις ουσίες. Αλλά εκεί όπως και αλλού, όπως προτείνει άλλωστε ο κύριος Ρολό, έχουμε συμφέρον να επιβάλλουμε την αρχή της πρόληψης. Αυτή η αρχή θα πρέπει να καθοδηγεί το κείμενο, η έκθεση στο, στο και στη φορμαλδεΐδη και άλλες ουσίες και στους πολυκυκλούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες πρέπει να επανεξεταστούν, όπως ζητεί και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Τέλος, να μην λησμονούμε και το ιατρικό προσωπικό που εκτίθεται σε κινδύνους ε, καρκίνου, γιατί εκτίθεται σε ουσίες μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες και σε φάρμακα ε, που καταστρέφουν τα κύτταρα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ρολάν που υποστηρίζει αυτή την αρχή της πρόληψης. Τη διατυπώνει επισήμως στην τροπολογία του παριθμού 18 και ότι υπενθυμίζει ότι πρέπει τακτικά να αναθεωρείται το κείμενο ούτω ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά ε, την άποψη των ιατρών, των ερευνητών, των επαγγελματικών συνδικάτων του τομέα της υγείας που αντιλαμβάνονται την ύπαρξη κινδύνων. Συμφωνώ απόλυτα με την επιμονή του να τονίζει την πρόληψη και να τονίζει και την ανάγκη ελέγχων. Τέλος, θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο να προσθεθεί μία αναφορά σε μελλοντικέ εργασίες όσον αφορά τις τοξικές ουσίες, ε, ανάδρομες τοξικές ουσίες, που είναι κάτι που επηρεάζει το ανθρώπινο είδος και θα πρέπει να υπάρξουν δομές παρακολουθής ιατρικής των εργαζομένων, κυρίως ε, η Επιτροπή Υγείας, οι γιατροί στον τόπο εργασίας, διότι χωρίς την προσπάθεια εκείνων δεν μπορεί να εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα. Ας επισημοποιήσουμε αυτό, αυτή την προσέγγιση μέσω τροπολογίας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καρή Μαντέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Ρολά. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε, λέει κυρία Ντέλη. Θα τα πω απλά τα πράγματα. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Βρισκόμαστε στην καρδιά του θέματος. Όταν μιλάτε για τις εκπομπές από τις κινητήρες diesel Κύριε Σιγητά, διορθώνεται το αξιοθρύνητο κενό και έλλειψη πολιτικού θάρρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτοντας εκπομπές που συνδέονται με το ντίζελ στο παράρτημα παριθμών 1, εκπομπές που είχε αφήσει εκτός προτάσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα των Πρασίνων, εν ονόματί μου ήδη είχε καταθέσει σειρά τροπολογιών σχετικών από την πρώτη φάση των συζητήσεων του κειμένου χωρίς να το μετανιώνουμε, λέω αυτό που λέω. Δεν λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μήνυμα που στέλνει. Αυτό θα έλεγα. Το Ευρωκοινοβούλιο αφιέρωσε μια ολόκληρη έρευνα όσον αφορά το Dieselgate. Θα περιμέναμε να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να αναφέρει στην έκθεσή τη τουλάχιστον το Diesel. Αυτό το κάνετε εσείς κύριε Σιγητά και σας συγχαίρω. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κατανοήσει πραγματικά, να καταλάβει αυτά τα στοιχεία που παρατίθενται. Πρέπει, είναι φρικτό, παίζουμε ακόμα με τα νούμερα, αλλά κάθε χρόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε Ευρωπαίος και κάθε Ευρωπαία εκτίθενται σε ρήπανση που προέρχεται από το ντίζελ. Τα είπε και ο κ. Λεγιαρίκ. 19 εκατομμύρια άνθρωποι, εργαζόμενοι, όλο και περισσότερο εκτίθενται λόγω επαγγέλματος της ουσίας. Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ταξινόμησε το ντίζελ στην κατηγορία των καρκινογόνων. Είναι σίγουρο, δεν είναι πιθανό. Πολύ πιθανό είναι σίγουρο. Ακόμα και χτες, βλέποντας τον τύπο, κυρίως τον γαλλόφωνο τύπο, που αποκάλυψε ένα καινούριο σκάνδαλο που συνδέεται με το Dieselgate. Αυτή τη φορά αφορούσε την Fiat Chrysler και επιβεβαιώνεται ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι μισθωτοί, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια θέση όσον αφορά τα ψέματα για το Diesel. Αλλά, άρα εκτιθέμεθα και στον επικίνδυνο χαρακτήρα της ουσίας. Το να συνδέονται στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας οι από το Diesel είναι το ελάχιστο δυνατό. Και δεν καταλαβαίνω πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξυπνήσει. Περιμένετε τι δηλαδή. Ένα δράμα όπως με, το, με, το, με τον αμίαντο. Τι περιμένετε εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν κύριε Σιγητά, αληθεύει ότι το δίζελ είναι το ελάχιστο δυνατό μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το εκρηκτικό κοκτέιλ που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα, έτσι. Στις νέες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να επομιστεί τις ευθύνες που έχει σαν νομοθέτης. Και γι' αυτό το λόγο θα υποβάλουμε τροπολογίες που θα επιτρέψουν να δράσουμε αμελητή όσον αφορά τοξική ουσία που έχει ταξινομηθεί το τρόπος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Προϊόντων, η Μπισφενόλη ε, Α. Άλλη τροπολογία. Να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των κινδυνευόντων πληθυσμών, κυρίως τις γυναίκες σε ηλικία αναπαραγωγής, τις εγγύους και την προστασία των εμβρίων πρέπει να λάβουμε υπόψη. Θα προτείνουμε ευθυγράμμιση των σχετικών μέτρων και των ορίων εκθέσεως βάσει των βελτίστων πρακτικών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει και για το ντίζελ. Η Ολλανδία προστατεύει καλύτερα από τη Γερμανία αντίθετα από αυτό που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του εισηγητού. Τέλος. Πρέπει να σας πω κύριε εισηγητά ότι αυτή η έκθεση δεν είναι κάτι αμεληταίο αν θέλετε πραγματικά η Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, να ξαναδώσουν εμπιστοσύνη, ξαναδημιουργήσουν εμπιστοσύνη σε μια Ευρώπη που προστατεύει, τότε πραγματικά θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες όσον αφορά την προστασία της υγείας. Να πληρώνουμε ένα μισθό σήμερα σε ένα μισθωτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε δικαίωμα στον εργοδότη να ρηπαίνει το μισθωτό. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν, να έχουμε υπόψη. Υπάρχουν τεχνολογικές βελτιώσεις σίγουρα, αλλά δεν πρέπει να έτσι ξαφνικά να αφήνουμε εκτός την αρχή της πρόληψης διότι είναι θέμα της υγείας των ανθρώπων που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και οι άνθρωποι δεν είναι πειραματόζωα. Αφού εργάστηκαν, επεξεργαζόμενοι, εκτιθέμενοι για 10, 20 χρόνια, 30 χρόνια σε χημικές ουσίες, δεν μπορούν να μπουν στη σύνταξη και να λένε έχω μόνο 5-10 χρόνια να ζήσω, διότι εργάστηκα σε συνθήκες που δεν είναι αξιοπρεπείς, με χημικά προϊόντα που δεν επιτρέπουν να ε, εκμεταλλευτώ τη σύνταξή μου. Αυτό θέλει να το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι σας διαβεβαιώνω ότι όσον αφορά το ντίζελ είμαστε στην αρχή της μάχης και δεν θα μας κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν μας αφήσει, δεν μας αφήσει, μα δεν μας κάνει κανείς ό,τι θέλει. Ευχαριστώ κύριε Ρολά. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος από το EFDD που θέλει να πει κάτι. Όχι. Άρα η κυρία Μελέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ρόλαν για την έκθεσή του. Δύο σχόλια έχω. Επί του τύπου καταρχάς. Πέντε επιτροπές ε, θα συμμετείχαν ε, στην ε, συνεργασία οι τέσσερις δεν συμμετείχαν η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας μου επέτρεψε να είμαι εισηγήτρια επί του θέματος για δεύτερη φορά η έκθεσή μου απορρίφθηκε, αφήθηκε εκτός υπό συνθήκες άκρως αντιδημοκρατικές πολύ κρίμα διότι πρόκειται περί συμπληρωματικότητας είναι σημαντικό αυτό και πάνω απ' όλα διότι στην πρώτη μου έκθεση σαφώς είχα υποβάλει το σοφώς στην αρχή της πρόληψης και στοιχεία προλήψεως όσον αφορά τα μόρια που σήμερα βρίσκονται σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή του κειμένου. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται γελία και θα ήταν γελία δεν ήταν το σοβαρό το θέμα. Επί της ουσίας η κατάσταση είναι σοβαρότατη. Και εκπλήσωμε διότι μιλάμε τόσο πολύ για τον ντίζελ ενώ όλες οι καρκινογόνες ουσίες δημιουργούν επαγγελματικούς ε, καρκίνους σε πολλούς κλάδους, δημιουργούνται αυτοί οι καρκίνοι και προφανώς θα πληρώσουμε με την υγεία των ανθρώπων. Μετά από περίπου 50 χρόνια όπου ήταν μετριοπαθής ο σεβασμός των κανόνων από πλευράς επιχειρήσεων. Λέμε σήμερα ότι υπάρχουν ελάχιστες τιμές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεννοούμεθα επ' αυτού. Αν αυτές οι οριακές τιμές είναι δύσκολο να γίνουν σεβαστές, δεν γίνονται σεβαστές, αυτό συμβαίνει και πρέπει να διαλέξουμε. Είτε οι εργαζόμενοι προστατεύονται όπως πριν ή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν. Εάν δεν υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι, δεν θα έχουμε ιδιαίτερη πρόοδο στο θέμα και κυρίως αν οι επιχειρήσεις παραβιάζουν τους κανόνες, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν συμπληρωματικό πρόβλημα. Δηλαδή, δύσκολο να απολαμβάνουν τους κόπους τους ε, διότι υπάρχουν διάφορες ουσίες που τους ρηπαίνουν, τρόποι μόλυνσης και διαφορετικές ε, χώρες όσον αφορά. Και αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών θα είναι πραγματική προσοκεφαλιά. Προσθέστε και, και λοιπά και το ότι δεν συμμορφώνονται οι, εργαζο... οι εργοδότες Πολύ λίγοι τελικά εργαζόμενοι που έχουν πληγεί θα μπορούν τελικά να καλυφθούν από την πρόνοια. Το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει όλα τα, τα μόρια τα καρκινογόνα να καλυφθούν και το ντίζελ, αλλά υπό συνθήκε που θα μπορούν να καλυφθούν είναι πολύ διαδεδομένη τοξική ουσία. Δεν αφορά μόνο μερικές εκθέσεις και υπάρχουν εκθέσεις στην ουσία εκτός επαγγελματικής ζωής. Και εκεί θα έχουμε προβλήματα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα, εάν κάνουμε πολλά πολύ γρήγορα κινδυνεύουμε να μην προστατεύσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε τον κύριο Λονά αποτελεσματικά σε κάτι ατμόσφαιρα και θα προσπαθήσουμε να είμαστε πραγματιστές όσον αφορά την προσέγγιση μας στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ρολά. Έξοχο το σχέδιο εκθέσεώ σας. Βασίζεται στα επιτεύγματά σας κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα τροπολογιών που αφορούσαν την οδηγία. θα έλεγα ότι είναι πολύ ισχυρή οδηγία. Η διαδικασία είναι κάπως δίσκαμπτη, αλλά συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιστήμονες, τα κράτη-μέλη, ε, καθ' τη διάρκεια της διαδικασίας. Έχουμε τέσσερα στάδια. Πρώτα απ' όλα έχουμε συνομιλίες του κοινωνικού εταίρους, μετά έχουμε επιστημονικές συμβουλές, μετά έχουμε τριμερή διάλογο, αξιολόγηση συνεπιών και μετά νομική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά υποβάλλεται η πρόταση. Όπως είδαμε και στην πρώτη αναθεώρηση που πρέπει να εγκριθεί. Έχει εγκριθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα προβεί στην έγκρισή του σε μια εβδομάδα πιστεύω. Στη διαδικασία αυτή με τα χαράς βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο σεβάστηκε τη διαδικασία. Και από το σχέδιο εκθέσεως του κ. Ρολαού βλέπουμε ότι έχουν επιτευχθεί ήδη αρκετέ βελτιώσει όσον αφορά την περιγραφή τη διαδικασία. Άκρο χρήσιμο αυτό. Οι στόχοι μας ποιοι είναι. επενδύουμε πόρους, πρέπει να κινηθούμε σωστά, άρα καλύπτουμε ομάδες ουσιών. Δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλους ταυτόχρονα, διότι πρέπει να γίνει σοβαρή αξιολόγηση. Είναι μια συνεχής διαργασία. Είναι σημαντικό για να απαντήσουμε στι ανησυχίε που εκφράστηκαν ότι πρέπει να μπουν περισσότερε ουσίε, ότι αυτό θα το κάνουμε σταδιακά. Οδηγία και αποτελέσματα. Ποιο είναι το σημαντικό. Πρέπει να δούμε ότι όταν συμπεριλαμβάνουμε μία ουσία στην οδηγία, όπως κάνατε και στα πλαίσια της προηγούμενης εκθέσεως για ε, τη σιλικόνη, την κρυσταλλική, την εισπνεόμενη, πρέπει να αντικατασταθεί ουσία καταρχάς. Η, η οδηγία δεν κάνει συμβιβασμού. Αν συμπεριλαμβάνεται μια ουσία, αυτομάτω αυτή πρέπει να αντικατασταθεί από άλλη ουσία από πλευρά του εργοδότου. Άρα, χρειάζεται σοβαρότατη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε, μπορούμε να προσμετρήσουμε την ουσία, τις συνέπειες κλπ. Αυτό το σεβαστήκατε και στην πρώτη έκθεση αλλά και στη δεύτερη. Όσον αφορά συγκεκριμένε ουσίε εκτιμούμε την πολύ ακριβή ε, περιγραφή της δραστηριότητας, αυτό είναι πολύ καλό και πηγαίνοντας στο diesel είναι σημαντικό να σημειώσεις Η Επιτροπή Σκολ έχει πάρει δημόσια θέσεις και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να τις υλοποιήσει κανείς, αλλά είναι όλα δημόσια αυτά, δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες παρερμηνίας. Υπάρχει επιστημονική συμβουλή να παραμείνουμε πιστοί στα πρότυπα των κινητήρων. Και όλες οι τεκμηριώσεις, όλη η συζήτηση που έλαβε χώρα με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων έχει αυτό τον περιορισμό, αν θέλετε. Η Επιτροπή, λοιπόν, θα υποβάλει με μορφή οδηγίας κάποιες προτάσεις, αλλά δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να υποβάλουμε τιμές που να, στο κείμενο αυτό που να ε, λαμβάνουν υπόψη και να τηρούν όλους αυτούς τους τύπους των κινητήρων. Βεβαίως και θέλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο θα συνεργαστούμε περαιτέρω μαζί σας. Απλώς ήθελα να σας επαναλάβω ότι η Επίτροπος Τίσεν, η Επιτροπή, είναι αποφασισμένη να πάρει πολύ σοβαρές δεσμεύσεις. Συμφωνούμε απολύτως με το σκεπτικό σας και θεωρούμε ότι η έκθεσή σας πραγματικά είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη. Πρόεδρος. Ο κύριος Ρελόν θέλει κάτι να πει. Πολύ σύντομα. Είναι εύκολο αν θέλετε το θέμα αυτό γιατί καμία πολιτική ομάδα δεν έχει διαφορετικές απόψεις. Όλοι θέλουμε να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αλλά να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Βέβαια είναι πιο περίπλοκο το θέμα από αυτό, γιατί υπάρχει και όλο το τεχνικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να το ε, αγνοήσουμε, να το εξαλείψουμε. Βεβαίως και η καπνή δίζελ είναι ένα από τα σημαντικά θέματα, καθότι αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους εγώ αποφάσισα σεβόμενος τις διάφορες γνώμες και την επιστημονική γνωμοδότηση και τις μελέτες να επιλέξω τον άνθρακα. Βεβαίως και υπάρχουν νέες τεχνολογίες και πραγματικά αν οι νέοι κινητήρες δίζελ μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα πρότυπα και τους νέους περιορισμούς, τόσο το καλύτερο. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταλάβει ότι θέλουμε πολύ, πολύ πιο πολλά στοιχεία. Πρέπει να είμαστε μεθοδικοί, πρέπει να είμαστε σοβαροί και είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μόνιμη και συνεχής αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Γι' αυτό και δεν έχω προσθέσει πολλά σημεία, δεν έχω υποβάλει. Συνάντησα πάρα πολλούς εργαζόμενους, αλλά και από τον τομέα της υγείας. Υπάρχουν άτομα που περιθάλπουν, που θεραπεύουν κάποιους οι οποίοι πάσχουν από τον καρκίνο και οι ίδιοι, οι ίδιοι είναι εκτεθειμένοι σε καρκινογόνες ουσίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης δεν θα πρέπει να έχουν χαμηλότερα ε, επίπεδα προστασίας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να στηρίξουμε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτήν την νέα νομοθεσία. Η συνοδεία πάντως, δεν ξέρω ποιος το ανέφερε αυτό, εσύ νομίζω Καριμά, η στήριξη των εργαζόμενων οι οποίοι πολλές φορές αρρωσταίνουν αφού έχουν σταματήσει να εργάζονται. Εννοείται ότι το θέμα αυτό είναι βεβαίως κοινωνικό Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, ασθενειών, νεκρών. Όμως, όμως, αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι και το οικονομικό κομμάτι, ο οικονομικός αντίκτυπος όλου αυτού του ε, τομέα. Και φυσικά, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η συμφωνία ΝΕΠΣΗ είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε και θα πρέπει όλοι οι φορείς να ενσωματωθούν σε τέτοιου είδους ε, διαδικασίες προληπτικές. Με αυτόν τον τρόπο πολύ πιο εύκολα λύνουμε προβλήματα σε τομείς όπου οι επιχειρήσεις, εάν έχουν προβλέψει με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κάποια πράγματα, προτρέχουν και προετοιμάζουν την νομοθεσία. Η νομοθεσία δεν μπορεί εκ των υστέρων να ε, ρυθμίσει όλες αυτές τις πτυχές. Με μεγάλη χαρά λοιπόν και με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω όλα στα σχόλια της προτάσεις σας γιατί πραγματικά είναι μια νέα αρχή και όπως σας είπα οι αναθεωρήσεις δεν θα σταματήσουν, θα είναι μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Εδώ και χρόνια στην Επιτροπή συζητάμε το θέμα αυτό. Αν θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταγωνιζόμαστε η μεν τους δε για χαμηλότερες καταβολές ποσών και για τις ίσες αμοιβέ, είτε πρέπει να συμφωνήσουμε αν θα υπάρξει μια κοινή αμοιβή για η διαργασία. Το θέμα τώρα της ε, έκθεσης σε καρκινογόνες ε, ουσίες νομίζω ότι είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ φιλόδοξα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων και κάποια άλλα κράτη-μέλη λιγότερο εκτίθενται εργαζόμενοι με άνισο τρόπο σε αυτές τις βλαβερές ε, ε, και καρκινογόνες ουσίες. Τώρα, 6 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Θα επεξεργαστούμε στις 22 και 23 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή της Επιτροπής 22-23 ε, Ιανουαρίου και ψηφοφορία 22 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Το επόμενο θέμα αφορά την απαλλαγή διάφορων ε, ιδρυμάτων. Κύριε Ρολά, έχετε το λόγο. Είστε εισηγητής και για το θέμα αυτό. Ναι, πραγματικά πιο απλό θέμα. Είναι οι γνωμοδοτήσεις για τις απαλλαγές για το 2016. Βασίστηκα στο, στις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα σας δώσω κάποια στοιχεία που θεωρώ σημαντικά. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει εγκρίνει τους ε, λογαριασμούς και των τεσσάρων αυτών ε, οργανισμών και Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά οι γνωμοδοτήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ενθαρρυντικές και υποστηρικτικές όσον αφορά την εργασία αυτών των ε, οργανισμών. Η εκτέλεση των προϋπολογισμών αυτών έγινε με υψηλά ποσοστά, με κάποιες μεταφορές ε, κονδυλίων κάτι το οποίο εδώ θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ αυτών των οργανισμών, συνέργειες ε, δημιουργούν και αυξάνεται η απατελεσματικότητά τους και αυτό είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω. Τρεις νομοθετικές ε, εκθέσεις όσον αφορά τους κανονισμούς τριών από αυτών των ε, οργανισμών, κάτι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, παραδείγματος χάριν. Υπήρξε πολύ σημαντική αναθεώρηση με καταπληκτική συνεργασία θα έλεγα και σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλους φορείς και οργανισμούς. Είναι σημαντικό επίσης να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η εκτέλεση των προϋπολογισμών έγινε με εξαιρετικό τρόπο και χαίρομαι ιδιαίτερα αγαπητοί φίλοι αν ε, με επικοδομητικό τρόμο μπορέσουμε να συζητήσουμε, αν έχετε παρατηρήσεις και σημεία, για τις γνωμοδοτήσεις μου, για τις απαλλαγές των διαφορών οργανισμών. Να ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, τον εισηγητή των σοσιαλιστών, ο κύριος Σάιμον έχει το λόγο. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να ανοίξω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, κύριε Ρολά. Για, για την εξαιρετική σας δουλειά. Όπως είπατε, και εμείς εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Όλα φαίνονται να έχουν εξελιχθεί ομαλά ε, κανονικά και νόμιμα. Πολύ σύντομα έχω κάποια σχόλια. Συμπληρωματικά με αυτά που είπε ο κύριος ε, Ρολά για το Eurofund φαίνεται ότι το Ίδρυμα αυτό λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο. Η ανάλωση των κονδυλίων είναι ε, εξαιρετική, σχεδόν 100%. Οι εκθέσεις τους, οι μελέτες τους, οι αναλύσεις τους είναι εξαιρετικές και πάρα πολύ χρήσιμες για μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Ο γενικός προϋπολογισμός τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 4,8% ε, σφάλματα για θέματα συνοχής ε, και εδαφικής ε, πολιτικής. Αυτό είναι υψηλό ποσοστό και συμφωνώ με την παράγραφο 4 του εισηγητή που λέει δεν χρειαζόμαστε επιπλέον μηχανισμούς ελέγχου αλλά καλύτερη εφαρμογή των υπαρχόντων μηχανισμών. Για το ETF, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήμουν ε, στο Τωρίνο πριν από λίγο καιρό για ένα γάμο και επισκέφτηκα τον ε, οργανισμό η το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρεται στα κτίρια αυτού του οργανισμού λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα και πιστεύω ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Πραγματικά λοιπόν αυτά τα ιδρύματα κάνουν εξαιρετική εργασία. Είναι χρήσιμα εδώ σε εμά την εργασία μας στο Κοινοβούλιο. Το βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο, 2015-2016, η εκτέλεση των προϋπολογισμών τους γίνεται με εξαιρετικό τρόπο, με υψηλά ποσοστά εκτέλεσης των κονδυλίων και η κατάσταση των Ιδρυμάτων αυτών είναι καλή και η έκθεση του εισηγητή εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάιμον. Η Ουλρίκε Τρεμπέσιος δεν είναι εδώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον από την ομάδα της. Άλτε. Ο κύριος Σελίμοβιτς για το γενικό προϋπολογισμό, το ETF και τα Ιδρύματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για την ε, πολύ ισχυρή του εργασία, τις εκθέσεις που μας παρουσιάζει τις γνωμοδοτήσεις για τις απαλλαγές. Βλέπουμε ότι αυτού του είδους ε, η γνωμοδότηση μας δείχνει πόσο καλή εκτέλεση του προεπολογισμού έχει γίνει από αυτά τα ιδρύματα. Στους περισσότερους τομείς που εξετάστηκαν, βλέπουμε ότι μπορούν να στηριχτούν μελλοντικέ προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό για μένα είναι προσυζήτηση, αλλά στο αφήσουμε προς το παρόν. Οι άλλες προτάσεις της Επιτροπής δεν θα πρέπει να συζητηθούν εδώ, αλλά κάπου αλλού. Εδώ μιλάμε μόνο για την απαλλαγή. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι κρίμα που τα θέματα που αφορούν την κοινωνική και δαυκή συνοχή για τις λιγότερο αναπτυγμένες επιτροπές χαρακτηρίζονται από πολλά σφάλματα, 4,8%. Αυτό το ποσοστό σφαλμάτων ξεπερνάει πραγματικά τα ανώτατα όρια και είναι ένα μαύρο σημείο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα λάθη αυτά γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Δηλαδή, μη επιλέξιμη ε, μη επιλέξιμα προγράμματα, μη επι, επιλέξιμα, σχέδια, κονδύλια και παραβιάσεις ε, των κανόνων και της νομοθεσίας που διέπουν τις προκήρυξεις διαγωνισμών Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρχει ένας τρόπος μέτρησης των αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων. Το 42% αυτών των προγραμμάτων δεν παρουσιάζουν τους στόχους. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός. Μετράμε όσον αφορά την εκτέλεση, την υλοποίηση, χωρίς να έχουμε το συγκεκριμένο ζητούμενο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει καλύτερος μηχανισμός για να ελεγχθεί αν έγινε βέλτιστη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και εδώ με πολύ ξεκάθαρο τρόπο οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αυξάνεται το γραφειοκρατικό άγχος, αλλά χρειάζονται διαδικασίες μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Θα αναφέρω λοιπόν εδώ ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός, καλύτερος έλεγχος και ιδιαίτερα όσον αφορά τον EFT, ETF, χρειάζεται βελτίωση όπως αναφέρει και το ελεγκτικό συνέδριο η κατάσταση των κτηρίων και οι 41 οργανισμοί, ιδρύματα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ε, έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου λειτουργούν ικανοποιητικά, αποτελεσματικά και είναι χρήσιμα. Είναι ουσιαστικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει έμφαση στην καλή διακυβέρνηση και στο τέλος του 2016 υπάρχει αύξηση του προσωπικού σε αυτές τις υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς σε σχέση με τα νούμερα του, των απασχολούμενων το 2015. Το θέμα του Brexit όταν αυξάνουμε τις αποστολές, το προσωπικό και μειώνουμε τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή. Επίσης θα πρέπει να μεταφερθούν και όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί και ιδρύματα που βρίσκονται στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή για τις ε, γνωμοδοτήσεις του και βεβαίως θα ακολουθήσει μια επικοδομητική συζήτηση. Η κυρία Έρκιν για τους υπόλοιπους ε, οργανισμούς και ιδρύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για τις γνωμοδοτήσεις του. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όπως είπατε, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους λογαριασμούς, είναι όλα νόμιμα και κανονικά και αυτό εξάλλου φαίνεται και από τις γνωμοδοτήσεις. Υψηλή ανάλωση των κονδυλίων και για τους τρεις αυτούς οργανισμούς και με αποτελεσματικό τρόπο. Για το Eurofound υπάρχει ένα θέμα με το καταστατικό του προσωπικού. Και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να συμπεριλάβουμε κάποια σχόλια γι' αυτό. Κάνω μια ερώτηση τώρα προς τον εισηγητή. Κάθε χρόνο, είτε είμαι σκιώδη εισηγητής, είτε είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες μεταφορές ποσών από το ένα χρόνο στο άλλο. Και άμα διαβάσει κανείς εκθέσεις καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά γιατί γίνονται για καλό σκοπό, για λογικό σκοπό. Αυτός ο ετήσιος χαρακτήρας κάποιων δαπανών Μήπως θα πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να αναγνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές, αν θέλουν να δουλέψουν καλά, πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να μην έχουμε κάθε χρόνο την ίδια πρόταση και την ίδια διατύπωση. Περισσότερη ευελιξία λοιπόν σε αυτό. Θα σε ευχαριστώ. Θα το σημειώσουμε αυτό και θα το συζητήσουμε όταν μπούμε στις λεπτομέρειες για τους οργανισμούς. Υπάρχει κάποιος που εκπροσωπεί τους πράσινους. Όχι. Την κουέ; Όχι. Η FDD δεν είχε σκιώδη. Η NF όχι. Από την Επιτροπή θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Όχι. Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τροπολογιών η υιοθέτηση 23 Ιανουαρίου 19 Μαρτίου στην επί Σαρμόδια επιτροπή και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης που είναι η παρουσίαση του εγγράφου εργασίας της ε, Επιτροπής κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Η κυρία Κάουφμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Να σας πω ποια είμαι. Είμαι διευθύντρια για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων στην ε, αρμόδια διεύθυνση υπεύθυνη για το συντονισμό του εξαμήνου, τον κοινωνικό διάλογο και είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας υποβάλλω με τους δύο συναδέλφους που είναι μαζί μου το θέμα αυτό που αφορά τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη. ΕΣΔΕ είναι τα αρχικά. Συνήθως το υποβάλαμε τέλος ε, του χρόνου, αλλά από φέτος ε, είναι έτοιμο το έγγραφο το καλοκαίρι, δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και αυτό βέβαια μας βοηθάει να αναλάβουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες και να έχουμε χρόνο μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Δημοσιεύουμε επίσης και μια άλλη έκθεση που αφορά την αγορά απασχόλησης, αγορά εργασίας, ε, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο και την ε, έκθεση για την απασχόληση χτες ε, παρουσιάστηκε αυτό και πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Συνήθως ε, έχουμε ένα θέμα, κυρίαρχο θέμα, και αυτή τη φορά αποφασίσαμε να μιλήσουμε για τις γενιές ε, και την ε, δικαιοσύνη μεταξύ γενεών ένα θέμα σημαντικό για όσους παίρνουν αποφάσεις για τις μελλοντικές ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα, αυτό το ΕΣΔΕ, τα θέματα των γενεών, συνήθως Ξεκινάμε με την παρουσίαση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε κάποιες βελτιώσεις. Φαντάζομαι ότι όσοι παρακολούθησαν το πακέτο για την απασχόληση που παρουσιάστηκε χτες θα το είδατε. Οι νέοι στην αγορά εργασίας, κοινωνικές συνθήκες ενσωμάτωσής τους, εντοπίζονται διαφορές αλλά και όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλά και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας τους υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται. Κοιτάμε επίσης λίγο και τη δημογραφική κατάσταση και υπάρχουν συνέπειες ιδιαίτερα αν κοιτάξει κανείς τη γύρανση του πληθυσμού είναι σημαντικό να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές γιατί βεβαίως θα πρέπει να δούμε ότι οι νέοι σε σχέση με τους ε, γυρεότερους βεβαίως ε, έχουν δυσκολότερη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας σήμερα, αλλά υπάρχει και το κόστος ε, της γενιάς αυτής που το αναλαμβάνει ε, η νεότερη γενιά, το κόστος περίθαλψης, το ότι σήμερα ζούμε πολύ περισσότερο. Αυτά επηρεάζουν την αγορά εργασίας την ίδια ώρα θα πρέπει να δούμε και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κατάσταση εδώ επιδεινώνεται. Βεβαίω έχουν αρχίσει να γίνονται μεταρρυθμίσει στον τομέα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και είναι προφανές μετά από όλα αυτά το που είπα το ότι χρειάζεται περισσότερη ενσωμάτωση εργαζομένων στην αγορά εργασία, περισσότερη παραγωγικότητα, ώστε να προσαρμοστεί η πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε. so, very... Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα είναι ότι είδαμε ότι το 2013 βελτίωση ε, της ε, απασχόλησης, μείωση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας τώρα είναι κατά μέσον όρο 7,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το 2008. Υπάρχουν βεβαίως σημαντικές αποκλίσεις. Βλέπετε ποια είναι τα σημεία απόκλησης και έχετε στα χειρότερα ποσοστά την Ελλάδα, στα καλύτερα την Τσεχία. Βλέπετε μεγάλες λοιπόν διακοιμάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η μακροχρόνια ανεργία επίσης έχει αλλάξει. Συγγνώμη λέει η μιλήτρια. Θα αλλάξω θέση. Όπως μπορείτε να δείτε ποια είναι η κοινωνική κατάσταση. Ε, σταθεροποιείται, υπάρχει και μια μικρή βελτίωση, κυρίως όσον αφορά το υψηλό ποσοστό το όχι όσον αφορά την εργασία, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση τα τρία τελευταία χρόνια. Υπάρχει όμως μία μικρή βελτίωση, παρόλα αυτά το ποσοστό φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού κάπως μειώνεται. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι επίσης Εάν συγκρίνουμε με τους ε, αριθμούς όταν αρχίσαμε και σήμερα, είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά. Στα πλαίσια της ε, στρατηγικής 2020 θέλαμε να έχουμε 20 εκατομμύρια λιγότερους φτωχούς στην Ευρώπη. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτό το θέμα της δικαιοσύνης μεταξύ των γενναίων. Βλέπετε ότι η τάση είναι ανωδική όσον αφορά το επίπεδο ζωής και την ευημερία. Πάντα πιστεύαμε ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, ότι οι νέοι θα ζουν καλύτερα από ότι εμείς. Αλλά είναι σαφές. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη αυτή την ανωδική τάση η κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά κυρίως τους νέους. Και η Λευκή Βίβλος του Μαρτίου αναφέρει ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι κάποιοι νέοι θα ζήσουν ίσως χειρότερα από ό,τι οι γονείς τους. Και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Γιούγκερ ανέφερε πόσο τον ανησυχεί αυτό για τις νέες γενιές. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ένα κλίμα δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Δεν είναι μόνο ο αντίκτυπο της κρίση μεταξύ των νέων που πρέπει να εξεταστεί. Ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργία μεταξύ των νέων, αλλά υπάρχει και το θέμα το δημογραφικό και πώς επηρεάζει την δυσαναλογία μεταξύ των νέων. Όλα αυτά όμως ξεπερνούν το τι πρέπει να γίνει για τους ε, νέους. Αλλά αυτό αφορά και το ΑΕΠ και όλα άλλα θέματα που επηρεάζουν τις ε, χώρες και την κοινωνική ανάπτυξη και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί σε επίπεδο ένωσης. Τώρα θα σας δώσω κάποια στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς ε, εργασίας και τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Θα δώσω όμως την δυνατότητα στον συνάδελφο να χειριστεί το κομπιούτερ γιατί εγώ δεν τα πάω καλά. Είπαμε. ότι στην αγορά εργασίας οι νέοι είναι αυτοί που υπέφεραν περισσότερο από την ενεργεία. Τα ποσοστά τους είναι ε, υψηλά και μετά από την ε, μείωση της ενεργείας στη δεκαετία του 90 τώρα έχουν αυξηθεί τα ποσοστά ενεργείας μεταξύ όλων των εργαζομένων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται λοιπόν για μεγάλη πρόκληση για τους νέους, όχι μόνο όσον αφορά τα εισοδήματά τους και την ε, πρόσβασή τους στην αγορά εργασία, αλλά το ότι δεν μπορούν να εργαστούν και να ε, εξειδικευτούν στην αγορά εργασίας για να έχουν ένα όπλο περισσότερο στα χέρια τους αύριο ψάχνοντας για εργασία. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερος κατακαιρματισμός όσον αφορά τη σταδιοδρομία των, των νέων οι εργαζόμενοι από 25 έως 9 ε, ετών είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, άτομα τα οποία όλο και λιγότερο όταν είναι νέα εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη περισσότερο ή έως 10 χρόνια. Πράγμα το οποίο προσθέτει στην ανασφάλειά τους. Ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι εργάζονταν ίσω όλη τη ζωή για τον ίδιο εργοδότη. Ναι. Είναι πιο εξειδικευμένοι οι νέοι, αλλά δεν έχουν τι ίδιες δυνατότητες στην αγορά. Και βεβαίως υπάρχει κάποιο το οποίο λέγεται non-standard work. Δηλαδή δεν κάνουν μία σταθερή εργασία σε μια επιχείρηση οι νέοι ή στην απασχόληση. Πολλές φορές δεν υπάρχει πλήρης απασχόληση και με οι νέοι αναγκάζονται να εργαστούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης με πρόσκαιρες συνθήκες εργασίας. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα λοιπόν για τους νέους. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει όσον αφορά την κοινωνική, τον κοινωνικό εστό των κοινωνιών. Επίσης, πρόσκαιρες συνθήκες εργασίας, προσωρινές συμβάσεις εργασίας, μειωμένα έσοδα και έτσι μεγαλύτερη συνεισφορά στα δημοσιονομικά και λιγότερα χρήματα στα συνταξιδοτικά συστήματα είναι τα επακόλουθα αυτής της κατάστασης. Τελευταίο θέμα που θέλω να σας παρουσιάσω, εν συντομία. Οι δημογραφικές εξελίξεις, βλέποντας πώς διαγράφεται το μέλλον. Βλέπουμε ότι πολλά άτομα δεν είναι πλήρως ενταγμένα στην αγορά εργασίας. Και βλέπουμε μείωση των ατόμων που είναι ενταγμένα στην αγορά εργασίας. Οι πρώτες που πλήττονται είναι οι γυναίκες Και αν κάνουμε συγκρίσεις με την αγορά τον ΗΠΑ, στην οποία υπάρχει αύξηση της ενσωμάτωσης των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, εμείς έχουμε μείωση. Επίσης, ε, γυράσκει ο πληθυσμός, δεν έχουμε πάρα πολλές γεννήσεις και αυτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στην αδελφό μου, την Αλέσια. Hi everybody. So after... Μετά από αυτή την ωραία ε, γενική επισκόπηση της έκθεσης θα ήθελα περισσότερο να αναφερθώ στα θέματα των ε, διαφορετικών γενεών στην αγορά εργασία και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τους νεότερους. Επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι στην αγορά εργασίας βλέπουμε πολλούς τρόπους αυτή τη διαφορά μεταξύ των γενεών. Είδαμε προηγουμένως έναν πίνακα στον οποίο φερόταν, φαινόταν η αύξηση ε, του, της ψαλίδας μεταξύ των γενεών. Είδαμε Τώρα, ανάλογα με τις ε, ηλικίε ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά εδώ δεν συμπεριλαμβάνουμε πάρα πολύ τους ε, νέους. Τι βλέπουμε, ότι σήμερα οι νέοι στην πράσινη γραμμή ακολουθούν ίδια ποσοστά και με την επόμενη ηλικιακή ομάδα, 40-64. αν και για αυτή την ηλικιακή ομάδα τα πράγματα βελτιώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση είναι οι νέοι, 25 με 3 νέα. Και τα ποσοστά απασχόλησης για αυτούς ε, μειώθηκαν περισσότερο. Επίσης, βλέπουμε ότι οι νεότεροι πρέπει να αντιμετωπίσουν στην αγορά εργασίας μεγαλύτερες προκλήσεις προκλήσεις που αντικατοπρίζουν και ε, δομικές ε, δυσκολίες και τις δυσκολίες που άπτονται της κρίσεις. Βλέπουμε ποια είναι η δύσκολη επαγγελματική κατάσταση για τους νέους. Το ότι δεν ε, καλύπτονται από τις συνήθεις και κλασικές συμβάσεις εργασίας. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν ε, προσωρινές συμβάσεις, προσωρινές συμβάσεις μερικής απασχόλησης και προσωρινές ε, συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Βλέπετε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του 2005-2016 για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν αυξήθηκε το ποσοστό εργασίας με κάπως ιδιότυπες συνθήκες εργασίας και αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι το ποσοστό των ε, ατόμων που εργάζονται με τέτοιου είδους συμβάσεις ε, είναι διπλάσιο όταν μιλούμε για τους νεότερους. Δείτε ποιες είναι οι διαφορές ε, λοιπόν μεταξύ της μπλε και της κίτρινης γραμμής. Τώρα δεν βλέπουμε στον πίνακα αυτά, αλλά βλέπουμε από μαρτυρίες ότι όπως προαναφέρθηκε το ποσοστό των νέων που εθελουσίως εργάζονται με συμβάσει μερικής απασχόλησης είναι πάρα πολύ υψηλό. Και οι προσωρινές συμβάσεις επίσης ε, ακολουθούν το ίδια ποσοστά. Βεβαίω όλοι θέλουν για να βελτιώσουν την εξειδίκευσή τους και για να έχουν μια κάποια σύμβαση μετά, ε, συγγνώμη, να έχουν στα βιογραφικό τους μια κάποια εμπειρία, δέχονται εθελοντικά τέτοιου είδους συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά. Οι μη συμβατικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι προβληματικές αφ' αυτού αλλά μόνο όταν συνδέονται κυρίως με πολύ χαμηλές αμοιβέ. Αυτό είναι το πρόβλημα, πολύ χαμηλές αμοιβέ. Στην πλεγραμμή βλέπετε το ποσοστό των εργαζομένων που έχουν ε, τις ε, συνήθεις πλήρους απασχόλησης και ε, α, αορίστου απασχόληση συμβάσεις, αλλά με χαμηλούς μισθούς. Επίσης, το πράσινο ποσοστό είναι μη συνήθεις συμβάσεις και χαμηλές απολαβές. Εδώ συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία έχουν πρόσκαιρες συνθήκες εργασίας. Και το σύνολο των δύο αριθμών βλέπετε ποιες είναι οι συνθήκες που Ακολουθούνται και οι εξελίξεις από το 2007 μέχρι σήμερα ανάλογα με τις ε, ηλικιακέ ομάδες. Βλέπετε λοιπόν ότι οι νεότεροι είναι αυτοί οι οποίοι ακτίθενται περισσότερο σε κακές συνθήκες εργασίας και κυρίως σε χαμηλότερες αποδοχές. Αυξήθηκαν οι πρόσχερες συνθήκες εργασίας και οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας για όλες τις ηλικιακέ ομάδες και η αύξηση ε, των ποσοστών αυτών σημαίνει ότι αυξήθηκαν και οι κακές αποδοχές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι νεότεροι είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από αυτές τις συνθήκες, αλλά τα άτομα γενικότερα που ε, υποφέρουν από αυτή το, και από μη συμβατικές συμβάσεις και από χαμηλές αποδοχές είναι αρκετά υψηλά. Αυτό είναι, ε, ναι, τη συγχωρείτε, αρκετά χαμηλά. Αυτό είναι θετικό μήνυμα μέσα στην κακή εικόνα. Τώρα βλέπετε ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτές τις συνθήκες για τους νέους στην αγορά εργασία το ότι είναι πιο εκτεθειμένοι σε μη συμφατικές συνθήκες εργασίας και χαμηλές αποδοχές οι νέοι, σημαίνει ότι τα μερίδιό τους στην, στα έσοδα και το, είναι οι μικρότεροι. Έτσι διαγράφονται οι τάσεις. Αν δείτε την τάση που αφορά τους νέους στο πράσινο κομμάτι, βλέπετε ότι μειώνεται η... το ποσοστό συνεισφοράς τους. Αυτό οφείλεται και στον αριθμό των εργαζομένων και για τη μέση αποδοχή ένα εργαζόμενο και αυτό για δημογραφικούς λόγους στον προηγούμενο πίνακα. Μία άλλη επίπτωση αυτής της κατάστασης δηλαδή οι επιπτώσεις για να παντρευτεί κανείς, να ανοίξει σπίτι. Παντρεύεται αργότερα, κάνει παιδιά αργότερα. Και έχει ερωτηματικά. Να περάσω σε αυτό το στάδιο. Βεβαίως, οι νέοι έχουν λιγότερες υποχρεώσεις όσον αφορά τις οικιακές δαπάνες. Αλλά Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και κάποια πράγματα. Όλο και αργότερα φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους οι νέοι, όλο και περισσότερο συγκατοικούν με άλλους νέους. Αλλά βεβαίως υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιο άλλο αποτέλεσμα είναι ότι αυξήθηκε ο μέση ηλικία των γυναικών όσον αφορά το πρώτο τους παιδί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, τα άτομα τα οποία σε ένα νέο νοικοκυριό είναι αυτά τα οποία ε, έχουν την κύρια απολαβή, ε, αυξάνονται, όσον, ε, ε, η ηλικία των ατόμων που σε ένα νοικοκυριό, νέο νοικοκυριό κερδίζει χρήματα αυξάνεται. Όλα αυτά λοιπόν τι μας δείχνουν. Ότι εκτίθενται περισσότερο σε τέτοιου είδους συνθήκες εργασίας ε, πρόσκαιρες οι νέοι. και βλέπετε ποια είναι το ποσοστό αυτών που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, πώς αυξάνεται, επαναλαμβάνω, η ηλικία της γυναίκες στην οποία θα κάνει το πρώτο του παιδί. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως απασχολεί και τους γονείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί την ε, κοινωνία όσον αφορά την ε, γεννητικότητα και κάτι το οποίο απασχολεί και τις κοινωνίες όσον αφορά το συνταξιδοτικό. Θα δώσω τώρα το, το λόγο στον συνάδελφο Γιώργ για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε σε πολλά επίπεδα να ενεργήσουμε για την κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο. Ε, είναι σημαντική η εκπαίδευση και η εξειδίκευση όπως είδατε είναι χρονικά όλο και περισσότερο σημαντική η εκπαίδευση. Επίσης, εξαιτία των αλλαγών στην αγορά εργασίας, είναι όλο και περισσότερο σημαντική η εξειδίκευση. Η επανεξειδίκευση η αγορά δεξιοτήτων επίσης είναι όλο και περισσότερο σημαντική. βεβαίω έχουν οι νεότεροι όλο και περισσότερο κίνητρα για να επενδύσουν χρόνο και χρήμα να κάνουν μια νέα εξειδίκευση για να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης, το, από ποια οικογένεια προέρχεται κανείς είναι πολύ σημαντικό για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ένταξη στην σύγχρονη κοινωνία μας και οι τεχνολογικές αλλαγές επίσης είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την όλη κατάσταση. Δίνω το λόγο τώρα στον Γιώργο. Good morning. Um, Καλησπέρα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να επιτρέψουμε στις κοινωνίες μας ε, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή η δυσχερή θέση των νέων στην αγορά εργασία αιτιολογείται κάτι τέτοιο. Διότι υπάρχουν και οι μεγάλες δημογραφικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εδώ βλέπετε την ε, ηλικία των ε, ενεργά εργαζόμενων μεταξύ του πληθυσμού. Δηλαδή, ηλικίες από 20 έως 64. Μείωση. Η διαφορά μεταξύ κόκκινης και πράσινης γραμμής είναι το ποσοστό ανεργίας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η διαφορά μεταξύ της μαύρης και της κόκκινης ε, γραμμής. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, γύρω στα 70 εκατομμύρια μη ενεργά οικονομικοί άνθρωποι σήμερα. Και βεβαίως για να διασφαλίσει κανείς ε, ε, την απασχόληση θα πρέπει να εξετάσει τα ποσοστά ανεργίας. Βεβαίως υπάρχουν ε, κάποιες υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον των ενεργών πολιτών. Ένα από τα σενάρια που βλέπω για το μέλλον είναι το ποσοστό δραστηριότητας εργασιακής. Δεν θα αυξηθούν αυτά, δεν θα βελτιωθούν αυτά τα ποσοστά. Στο παρελθόν είχαμε σημαντικές αυξήσεις, αλλά δεν προβλέπεται περαιτέρω αύξηση. Τώρα, με το σενάριο υψηλής δραστηριότητες κάνω κάποιες υποθέσεις πάρα πολύ ε, και κάποια σενάρια, κάποια πολύ αισιόδοξα. Βεβαίω, η δραστηριότητα των ατόμων αυξάνεται ανάλογα και με το επίπεδο εκπαίδευσή τους. Αυτό όμως το αισιόδοξο σενάριο που βελτιώνεται σε ποστό 23% σημαίνει ότι όλοι θα είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας. Βλέπετε όμως ότι μιλάμε για 30 εκατομμύρια άτομα όταν μιλάμε μεταξύ του σενάριου υψηλής και Χαμηλή Γι' αυτό η πολιτική μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορέσουν να, να εισέλθουν στην αγορά πολύ περισσότερα άτομα στα πλαίσια αυτής της high activity. Πώς διαγράφεται η απασχόληση. Στο παρελθόν είχαμε ένα ποσοστό 1,1%. Ε, Βεβαίω τα ποσοστά αυτά διαψεύτηκαν μετά από την οικονομική κρίση και άλλαξαν. Από το 2013 λοιπόν και μετά βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξαναγυρίζουμε σε αυτά τα ποσοστά, τα 1,1%. Αν συνεχίσουμε με αυτά τα ποσοστά θα φτάσουμε στα ποσοστά τα οποία είχαμε προβλέψει μετά από πολλά χρόνια. Αρκετά αργότερα. Στο low activity σενάριο, αν δεν γίνουν περαιτέρω θετικές προσπάθειες, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι η περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης πολύ σύντομα θα σταματήσει να αυξάνεται και, κά... και αμέσως μετά το 2020 θα έχουμε αρνητική ε, και αν δεν μπορέσουμε να εντάξουμε στην αγορά εργασίας πολύ περισσότερα άτομα, αυτό το ποσοστό 1,1% θα αφορά μόνο ελάχιστα άτομα, άρα το 2030 θα βρισκόμαστε στην κατάσταση που σκεφτόμαστε ότι θα επικρατήσει το 2020. Ακόμη και αν κινητοποιήσουμε όλες τις, ε, τους δυνατούς πόρους που έχουμε για να ενεργοποιήσουμε την αγορά, η απασχόληση θα σταματήσει να αυξάνεται και θα αρχίσει να μειώνεται, διότι και το ηλικιακό φάσμα των εργαζομένων θα αρχίσει να, μιλών, να μειώνεται. Βλέπετε σε αυτό το πίνακα κάποιες δυνητικές αυξήσεις του ΑΕΠ της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Βλέπετε λοιπόν ότι από το 2 στο 2008 έτσι είχαν τα πράγματα από το 8 μέχρι το 13. Δεν θα αναφέρω στο διάγραμμα τι ακριβώς συνέβη. Από το 13 στο 16 βλέπουμε ότι η κατάσταση μοιάζει με αυτή που επικρατούσε από το 2000 μέχρι το 2008. Υπάρχει μια κάποια σταθεροποίηση αλλά σε χαμηλότερα ποσοστά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε για το μέλλον ότι η αύξηση του ΑΕΠ 2% είναι περίπου το σημείο ισορροπίας, είναι ο μέσος όρος. Τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αύξηση του ΑΕΠ σε ποσοστό 2% σε, 2, ε, σε ποσοστό 2%. Αλλά εάν στο μέλλον έχουμε ανάπτυξη μόνο 1,5%, τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα. Διότι η αύξηση της απασχόλησης θα είναι μειωμένη, άρα για να είμαστε στο ίδιο ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ θα πρέπει να βελτιώσουμε μαζικά την παραγωγικότητα. Αυτά στα πλαίσια του σενάριου Χαμηλή δραστηριότητα. Εάν έχουμε το άλλο σενάριο, το υψηλό, διαμορφώνονται έτσι με τα στικτά, ε, με στικτά διαστήματα οι εξελίξεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό της ε, ε, δικαιοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διαφόρων γενεών. Ξέρουμε ότι στην αγορά εργασίας και το επαναλαμβάνω οι νέοι βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση. Και σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το σενάριο, τι πρέπει να κάνουμε για την κατανομή του ΑΕΠ, για να είμαστε πιο δίκαιοι. Σκεφτείτε κάτι το διαφορετικό. Α σκεφτούμε ότι είναι μία χώρα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα συνταξιδοτικό σύστημα και όλοι από 20 μέχρι 65 εργαζόταν. Και όλοι πάνω από 65 ήταν συνταξιούχοι. Και ας πούμε ότι το επίπεδο των συντάξεων ήταν 47% τη μέση της μέσης αμοιβή. Εν τη αυτή περιπτώσει είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να υπολογίσει κανείς ότι χρειάζεται 14% του ποσοστού συνεισφοράς για το συνταξιωτικό σύστημα από τον εργό πληθυσμό για να εξισορροπήσει τα έσοδα με τις δαπάνες με το ρυθμό που κινείται το συνταξιωτικό σύστημα. 14% μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά τα επίπεδα παρόλη τη δημογραφική αλλαγή. Δεν το φαντάζομαι. Κοιτάξτε τη γαλάζια γραμμή που αναφέραμε, τη μείωση του πληθυσμού σε εργασία ηλικία και η κόκκινη γραμμή, η αύξηση του πληθυσμού που είναι σε ηλικία μεγαλύτερη από 65, του συνταξιούχου. Αν θέλουμε να παραμείνουν τα συνταξιωτικά επίπεδα 47% του μισθού, το ποσοστό της συνεισφορά θα πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί στο μέλλον. Εν τη απουσία άλλων μεταρρυθμίσεων. Και θα μπορούσε να πει κανεί καλώ δεν μπορούμε να διπλασιάσουμε τη συνεισφορά. Σκεφτείτε το κόστο εργασία, το εργατικό κόστο και τι αμοιβέ, τι καθαρέ. Δεν είναι δυνατόν. Δεν επιτρέπω να αυξηθεί καθόλου η συνεισφορά συνταξιδοτική, οπότε θα πρέπει να την πληρώσει τελικά η σύνταξη. Καλή τύχη στους συνταξιούχους. Τι θα γίνει στο μέλλον, λοιπόν. Κάτι ενδιάμεσο μεταξύ των δύο ακραίων ενδεχομένων. Είμαι σίγουρος, σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Στο μέλλον θα γίνει. Η δημογραφική αλλαγή μέσω της γύρανσης θα κάνει τον κόσμο, τους πολιτικούς να σκεφτούν ότι κάποια αύξηση στη συνεισφορά είναι αναπόφευκτη. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Θα πρέπει να μειωθεί, να συγκρατηθεί η αύξηση των συνεισφορών. Ή αυτό ή το εργατικό κόστος. Και ας πούμε ότι σταματάμε στο 20%. Δεν επιτρέπουμε τις συνεισφορές να αυξηθούν πέρα από το 20%. Γιατί αυτή αυτή περίπτωση το επίπεδο των συντάξεων, το κόκκινο, μπορεί να παραμείνει στο 47% στο βαθμό που το επίπεδο συνεισφοράς ε, μπορεί να αυξάνεται ελεύθερα. Εν τω μεταξύ, μειώνουμε το, κρατάμε, συγκρατούμε στο 20%, αρχίζουν να πληρώνουν οι συνταξιούχοι αποδεχόμενοι χαμηλότερες ε, συντάξεις. Το 2060-2070 ότι το κόστος της γύρανσης διαιρείται μεταξύ των εκείνων που θα συμβάλλουν στο μέλλον και εκείνων που θα είναι συνταξιούχοι. Οι μεν θα αποδεχτούν χαμηλότερε συνθήκε και οι δε θα πρέπει να αποδεχτούν μεγαλύτερε συνεισφορέ. Μπορεί να διερωτηθεί κανεί αν αυτό είναι δίκαιο. Αν είναι δίκαιο, αν θεωρηθεί δίκαιο, πρέ, πρέ, πρέπει να δούμε ε, κάποιου που γεννούνται μια χρονιά. Ξεκινάμε το 1997, του σημερινού νέου που μπαίνουν στην αγορά εργασία. Και τι βλέπετε, ότι οι σημερινοί νέοι σε όλη τη ζωή θα πληρώνουν κατά μέσο όρο πολύ ψηλότερη συνεισφορά από ό,τι είναι ο μέσος όρος σήμερα. Και εκείνοι οι ίδιοι ταυτόχρονα, όχι ταυτόχρονα, αργότερα, σαν συνταξιούχοι, θα πρέπει να έχουν μειωμένη σύνταξη, πολύ χαμηλότερες συντάξεις από ό,τι οι σημερινοί συνταξιούχοι. Διπλό βάρος της γύρανσης το αποκαλούμε αυτό. Ζητούμε από τους σημερινούς νέους, τις μελλοντικέ γενιές, το διπλό βάρος της γύρανσης να υπομισθούν. Και κλείνω άλλη μια διαφάνεια τι συμβαίνει αν όλοι εργαστούν άλλο ένα χρόνο. Ένα χρόνο παραπάνω. Βλέπετε τη διαφορά. Αν όλοι εργαστούν μόνο ένα χρόνο, χρόνο παραπάνω, τελικά ε, με την παρούσα εισφορά μπορούμε να έχουμε ψηλότερε συντάξει, πολύ ψηλότερε συντάξει. Άρα, ενεργοποίηση στην αγορά εργασία είναι μια απάντηση. Επένδυση στην απασχολησιμότητα των ανθρώπων. Και εδώ τελείωσα. Πρόεδρος, άλλο ένα λεπτό. Θα είμαι συντομότατη. Άλλο κεφάλαιο ασχολείται με τον κοινωνικό διάλογο και βλέπουμε ότι όταν οι νέοι δεν εκπροσωπούνται παρκώς τα συνδικάτα, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ότι αυτό είναι γεγονός και πιθανότατα να έχουν προσωρινή απασχόληση οι νέοι και όταν έχουν προσωρινή απασχόληση είναι μικρότερη συμμετοχή στη συνδικάτα και στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται τόσο πολύ από τις συλλογικέ συμβάσεις όσο οι πιο ηλικιωμένοι και αυτό εξαρτάται και από τον τομέα οπότε είναι και θέμα εκπροσώπησης των νεωτέρων εργαζομένων στα συνδικάτα και πρέπει να δούμε και την βελτίωση της εκπροσώπησής τους. Και στην άλλη σελίδα βλέπετε ότι υπάρχει κάποια δράση που δρομολογείται και από εργοδότες και από συνδικάτα προσπαθούν να το περισσότερο οι πιο νέοι και οι πιο ηλικιμένοι εργαζόμενοι. Υπάρχει και συμφωνία για την ενεργό γύρανση τα προβλήματα ήδη περιγράφησαν λεπτομερώς με την αγορά εργασίας, τα συνταξιωτικά συστήματα, θέματα αποφάσεων ζωής επίσης αναφέρθηκαν και πολλές από τις συστάσεις για την πολιτική, είτε είναι η πρωτοβουλία της δεξιότητες ή άλλη πρωτοβουλία, γίνονται προσπάθεια. Και η διακήρυξη του κοινωνικού πυλώνα έχει τεθεί επίσης. Άρα Όλα αυτά είναι σημαντικά, όχι μόνο για τη βελτίωση της συγκλήσεως μεταξύ κρατών μελών, αλλά και όσον αφορά την βελτίωση της κοινωνικής καταστάσεως εντός των κρατών μελών. Πρέπει να έχουμε υπόψη και κάποια, κάποιες πτυχές που συνδέουν τις διάφορες γενιές και αφορούν τη βελτίωση της καταστάσεως των νέων, τις προπτικές που έχουν οι νέοι, και το τι μπορούν να κάνουν οι διάφοροι θεσμοί, οι δημόσιοι για τη βελτίωση της καταστάσεως των νέων. Αυτά και σταματώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τις διαφάνειες που μας δείξατε, μήπως θα μπορούσαμε να τις έχουμε για να διανεμηθούν στα απουσιάζοντα μέλη, στα πόντα μέλη. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε τα ακριβή στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Αν κάποιος επιθυμεί να προβεί σε κάποιο σχόλιο, ελεύθερα. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, λέει ο κ. Γοσφό, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έκανε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τη χρειαζόμαστε. Πριν από την κρίση της, δεκα... της τελευταίας δεκαετίας το συζητούσαμε εκτενώς. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της κρίσεως εστιαστήκαμε επί των θεμάτων της κρίσεως ε, και λησμονήσαμε αυτά που συζητάμε σήμερα λίγο. Ε, δύο πτυχές σημαντικές παρουσιάστηκαν στις παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε γενικά την προσέγγιση που ακολουθείται την οικονομική. Τονίσατε κάποια πράγματα. Κάποια προβλήματα είχαν εμφανιστεί πριν από την κρίση. Η προσωρινή απασχόληση των νέων Φερρυπίν και η απασχόληση των πιο ηλικιωμένων ήταν κάτι που είχαμε ε, συζητήσει πριν από την ε, κρίση. Κάτι που είναι πιο εντυπωσιακό και συνοψίζει αυτά που είπατε. Σήμερα η γενιά που πληρώνει είναι η διάμεση. 35 με 55. Για να το πω απλά. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα έχουμε ξανά νέους, επειδή έχουν επισφαλή εργασία, πρέπει να συνεχίσουν να βοηθούνται από τους γονείς τους και συνταξιούχους που θα πρέπει να βοηθούνται αυτοί από τα παιδιά τους, διότι η σύνταξή τους θα μειωθεί και με τη μεγάλη ηλικία που έχουμε σήμερα, σε πολλές ηλικίες έχουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι 90-92 ετών που έχουν τις ασθένειες της γύρατος και πρέπει να βοηθηθούν και αυτοί από τις οικογένειές τους διότι το σύστημα δεν μπορεί να τους αναλάβει. Και την κατάσταση, ξέρουμε και θα γνωρίσουμε αύριο αφόρητες καταστάσεις που υπάρχουν μόνο μια δραστήρια γενιά που έχει πίσω της μια γενιά πιο νέα και μια πιο ηλικιωμένη που θα πρέπει εν μέρη να βοηθά τους άλλους από το μισθό τους. Το θέμα το σημαντικότερο είναι τι πρέπει να κάνουμε βέβαια. Από αυτά που είπατε το είδαμε. Συμφωνώ με τα συμπεράσματά σας. Τελικά να χρησιμοποιήσουμε μόνο την αύξηση των εισφορών δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να χρησιμοποιήσουμε μόνο την μείωση των συντάξεων δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν αναμίξουμε τα δύο δεν είναι ικανοποιητικό. Χρειαζόμαστε μείγμα πολιτικών. Οπότε γίνεται και θέμα, τίθεται το θέμα ηλικία συνταξιοδότησης. Μπορούμε συνεχώς να προωθούμε το έτος συνταξιοδότησης και να απασχολούμε τους ανθρώπους 60, στα 65 κλπ. Ρίξατε μια ιδέα να εργάζονται οι εργαζόμενοι ένα χρόνο παραπάνω. Εγώ πιστεύω σε αυτή τη λύση ε, και σαν φιλελεύθερος, επειδή πιστεύω ότι η δουλειά είναι κάτι θετικό, άρα μπορούμε να το προτείνουμε να το κάνουν οι άνθρωποι επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν βελτιώνται τις συνθήκες ζωής και αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Αλλά δεν γίνεται αυτό αυτόματα αν δεν αλλάξουμε τις συνθήκες εργασίας. Έκανα μελέτες επ' αυτού. Και πιστεύω ότι αν θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό δραστηριότητας των ανθρώπων που είναι 64, 65, 66 ετών, από 45 ετών πρέπει να ξεκινήσουμε την κατάρτιση των μισθωτών. Να δουν τι δραστηριότητες θα μπορέσουν να, να ασκήσουν όταν όταν 60-65. Να λέμε, το, στις δίσκος εργασίες εργαστήκατε μέχρι τα 62 και τώρα θα πρέπει να εργαστείτε μέχρι τα 65, αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι κάτι που κουράζει ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους. Και πάση περιπτώσει επιχειρήσεις δεν θεωρούν ότι είναι πλεονεκτικό, διότι η παραγωγικότητα, η ατομική αυτών των μισθωτών είναι πάρα πολύ μικρή. Να το πούμε αλλιώ, κλείνοντα. Δύο στοιχεία πρέπει να προωθηθούν. Ποιοτικού χαρακτήρα. Στην πρότασή σας. Το πρώτο στοιχείο. Το θέμα της κατάρτισης, το αναφέρατε. Εντός της καταρτήσεως είναι η διαβίου κατάρτισης που συμπεριλαμβάνεται. Όχι όταν είναι κάποιος 20-40, κατάρτιση και όταν είναι κανείς στα 45, στα 50, στα 55, όσον αφορά το είδος των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να εξασκηθούν όταν κάποιος είναι 64-65 ετών για να είναι πάντα χρήσιμος. Βέβαια θα υπάρχει και φθορά της ηλικία που είναι η κανονική φθορά ε, της παραγωγικής δυνατότητας που δεν είναι η ίδια για όλα τα επαγγέλματα, αλλά υπάρχει. Άλλη ποιοτική λύση. Για το τέλος ενεργού ζωής πρέπει να υπάρχει και μερική δραστηριότητα, όχι πλήρους απασχόλησης. Ίσως για ένα-δύο χρόνια ο χρόνος εργασίας να αυξηθεί με μερική απασχόληση. Εν τη αυτή η περιπτώση, ποια είναι η δυσκολία να έχουν τα δικαιώματα συνταξιοδότηση με μερική απασχόληση με αυτού που έχουν πλήρη απασχόληση. Αλλιώ δεν θα συνδεθούν με τη μερική απασχόληση ή θα αισθανθούν ότι θα χάσουν από τη σύνταξή του. Υπάρχουν διάφορα πράγματα λοιπόν προ ανάλυση και προβληματισμών. Δύσκολο να συνδεθούν, να συνδεθούν όλα αυτά. Και υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που έλειψε την παρουσίασή σας. Δεν ξέρω αν το έχετε λάβει υπόψη, πολύ σημαντικό. Το θέμα της μετανάστευσης. Εσείς κάνατε μια υπόθεση κλειστής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρόνια όμως που έρχονται θα είναι πολύ σημαντικός ο παράγων μετανάστευση. Ποιες θα είναι οι συνέπειες μετανάστευσης; Θα μειώσει τις διαφορές μεταξύ των ομάδων που παρουσιάσατε. Εγώ δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Τροφή προσκέψη λοιπόν. Για τις μελέτες σας που υπήρξαν άκουσαν ενδιαφέρουσες. Και όπως είπατε Πρόεδρε, περιμένω ανυπόμονα να τις δω γραπτές και να τις διαβάσω προσεκτικά. Τις μελέτες παρουσιάστηκαν προφορικά. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Χάρκιν. Και μετά θα σας αφήσω να προσπαθήσετε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσει Η κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έξοχη παρουσίαση. Κάπου αλλού έπρεπε να είμαι τώρα. Αλλά ήταν τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά που έπρεπε να μείνω και να ακούσω ο συνάδελφός μου ο κ. είπε τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω, με κάλυψε. Άρα δεν θα τα επαναλάβω. Συμφωνώ όμως ότι το θέμα αυτό κάπως ξέφυγε από το θεματολογιό μας. Είχαμε πολλά άλλα θέματα που μας απασχολούσαν. Και έτσι δεν ήταν αυτό το θέμα στο επίκεντρο όπως το αρμόζει. Τι πιστεύω εγώ. Υπέχουμε ευθύνη πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ασδήποτε λύσης που θα προταθεί, διότι εκπροσωπούν όλες τις γενιές. Σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την επικείμενη κρίση. Το μήνυμα πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο που δεν θα διχάσει τις γενιές και να μην αρχίσουν οι κατηγορίες των μεν κατά τον δε. Δεν βοηθάει κανέναν αυτό. Και θα μας οδηγήσει αυτό σε βιαστικές λύσεις που δεν θα είναι βιώσιμες και δεν θα είναι αποδοτικές. Η διπλή συνεισφορά η περικοπή των συντάξεων κατά το ίμιση ήταν σκοτεινά σημεία. Ακόμα και αυτά αν τα κάνουμε δεν αρκούν. Ίσως χρειάζεται να εργάζονται οι άνθρωποι παραπάνω. Και εξαρτώνται όλα αυτά από την προσαρμοστικότητα των αντόμων, από τον τόπο εργασίας κλπ. Μάλλον στραβά το πιάσαμε το ζήτημα. Γιατί το λέω αυτό. Οι νεότεροι έχουν άθελά τους μερική απασχόληση. Ίσως οι πιο ηλικιωμένοι θα έπρεπε να έχουν αυτή την ευκαιρία της μερικής απασχόλησης και οι νέοι να είναι εκείνοι οι οποίοι ίσως να έχουν πιθα... δυνατότητες πλήρους απασχόλησης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιστρέψουμε την προσέγγιση. Πρέπει να το δούμε όμως. Υπάρχει εντύπωση ότι όταν κάποιος φτάσει σε μια ηλικία πάνω από τα 60, ότι η σύνταξη είναι κάτι αυτόματο. Αυτό δεν ισχύει παντού. Εν γένει όμως αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτή την αντίληψη να την αλλάξουμε. Όχι λέγοντας απλώς στον κόσμο πρέπει να δουλέψετε μέχρι τα 67, μέχρι τα 68 ή μέχρι τα 69 σας ή οποιαδήποτε άλλη ηλικία. Πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα τέτοια που θα επιτρέπουν στον κόσμο να μειώσει, να απομακρυνθεί κάπως από την εργασία του αν αυτό επιθυμεί με τρόπο τέτοιο που ούτε τόσο ώστε να μην είναι μια απειλή που επικρέμεται πάνω από το κεφάλια. Θα είναι μια ευθύνη που αναλαμβάνει κάθε γενιά. Θα είναι πιο υπεύθυνη η προσέγγιση. Το τελευταίο σχόλιο ήταν εξίσου σημαντικό. Ποιο θα είναι ο αντίκτυπο τη μετανάστευση. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό γιατί το ερώτημα ήδη έχει τεθεί. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάφμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια. Για το θέμα της μετανάστευσης θα ζητήσω από τον Γιώργ να μπει στις λεπτομέρειες. Αναφέρεται στην έκθεση. Ξεκινά λοιπόν λέγοντας ότι είπατε ότι το ποσοστό απασχολησιμότητας ή δραστηριότητα των πιο ηλικιωμένων πριν από την κρίση ήταν αρκετά χαμηλό. Πράγματι. Έχουμε θετική εξέλιξη όμως σε αυτό. Το 2006 η απασχολησιμότητα των ηλικιωμένων εργαζομένων ήταν 43%. Τώρα είναι 55%. Άρα έχουμε μια συνεχή ανωδική τάση όσον αφορά τη συμμετοχή των πιο ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό. Πρέπει να συνεχιστεί. Συμφωνώ ότι το είδος της εργασίας έχει σημασία. Το πώς εργάζονται οι άνθρωποι. Τα κράτη-μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Δύσκολο εμείς να μετρήσουμε τις ώρες εργασίας, πόσο δουλεύουν οι πιο μεγάλοι σε σχέση με, πιο, τους πιο νέους κλπ. Σε ένα άριστο θέμα θα υπάρχει σταδιακή μείωση των ωρών. Διαβίω εκμάθηση. Σημαντικό θέμα. Όπως είπε ο Γιώργ, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και πρέπει να αυξηθεί για τους νέους. Είμαι πεισμένοι ότι πρέπει για όλους να αυξηθεί. Με άλλα λόγια, αν έχουμε διαβίω εκμάθηση, θα πρέπει και η παραγωγικότητα των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων να αυξηθεί. Άρα, διευκολύνεται η κατάσταση έτσι, παρά αν εστιαστούμε μόνο στους νέους για την αύξηση της παραγωγικότητας. Χρειαζόμαστε μία προσέγγιση κοινή σε όλα τα μέτωπα, σε όλες τις ηλικίες. Να στραφώ στις ώρες που αναφέρθηκαν. Τι παρατηρούμε Όσον αφορά την ανεργία, τα ποσοστά ανεργίας, είμαστε στα επίπεδα του 2008, αλλά όχι όσον αφορά τις ώρες εργασίας. Η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση είναι καλύτερη όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων από ό,τι όσον αφορά τις ώρες εργασίας. Είναι σημαντικές και ώρες εργασίας. Το είδα σε μια διάσκεψη αυτό. Όσον αφορά τις ανισότητες. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και κάτι άλλο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Να, μην κατηγορεί μια κατηγορία εργαζομένων τους άλλους, μια ηλικία τους άλλους. Θέλαμε να ρίξουμε φως στους νέους κυρίως, στην ανάλυση που κάνουμε, αλλά δεν πρέπει να κατηγορούμε το τρόπο στους ηλικιωμένους. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τους νέους τι πολιτικές χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τη μετανάστευση, να πω καταρχάς ότι η προηγούμενη έκθεση είχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στη μετανάστευση και πώς ανάλογα με τις δεξιότητες που έχουν ή το φίλο τους είναι καλύτερη ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας ή λιγότερο καλή. Είναι κάτι που εξετάζουμε εκ του στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εξετάζοντας κάθε χώρα, εκεί εστιαζόμαστε. Θέλουμε η ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό να είναι καλύτερη. Κατά την άποψή μας, αυτό ξεκινά από τη φροντίδα των παιδιών ήδη. Ξεκινά από τη βελτίωση των παιδιών που προέρχονται από μετανάστες κινητικότητα κοινωνική προς τα άνω. Επίσης, όσον αφορά τις προσωμείωσεις, μπορεί να εξηγήσει μια από αυτές ο Γιώργ καλύτερα. Εξετάζει το τι μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε το εργατικό δυναμικό και να το αυξήσουμε το εργατικό δυναμικό μέσω της καλύτερης ένταξης των μεταναστών ή ανθρώπων από, ε, που προέρχονται από περιβάλλον μεταναστευτικό. Το συμπέρασμά μας δεν είναι ότι πρέπει να εργάζονται όλοι ένα χρόνο παραπάνω. Κάναμε μια προσωμείωση για να δείξουμε τι θα γινόταν αν όλοι εργαζόμασταν ένα χρόνο παραπάνω. Αυτό είναι μια κατάσταση που ποικίλει από χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες είναι πιο προχωρημένες, άλλες πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα και το πού έγκυται η λύση είναι κάτι που θα είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης ανάλυσης. Ο Γιώργο, ευχαριστώ. Όπως είπε και η Μπάρμπαρα, αναφερθήκαμε στη μετανάστευση, στην έκθεσή μας. Παίξαμε κάπου με τις υποθέσεις που χρησιμοποίησαμε και τι συμπεράναμε, ε, ότι αν διπλασιάσει τα ποσοστά μετανάστευσης σήμερα, μέχρι το 2025, σταδιακή αύξηση, πάνω από μία δεκαετία, βελτιώνεται η κατάσταση. Μεσοπρόθεσμα θα μειώσεις την πίεση όσον αφορά την παραγωγικότητα, αλλά δεν θα εξαλειφθεί η πίεση της παραγωγικότητας τα επόμενα χρόνια θα είναι ε, σταθερή, σχετικά σταθερή. Σχετικά με αυτό. Αναφερόμενος στις περικοπές των συντάξεων. Τι κάνω σε αυτό το διάγραμμα. Κάποια ώρα το χέρι παίρνει από τους συνταξιούχους. Περικοπές. Κάνει περικοπές από τις συντάξεις. Δεν συμπεριλαμβάνω το διάγραμμα τη πιθανότητα ε, μεγαλύτερης μετανάστευσης και ε, μετάθεσης για μεγαλύτερη ηλικία του έτους συνταξιοδότησης. Χρειάζεται πολιτικό μείγμα. Πρέπει να έχουμε μελλοντική ανάπτυξη. Αυτή είναι μια πίεση. Και χρειάζεται ισολογισμός των συστημάτων των συνταξιδοτικών. Δεν μιλήσαμε για τη γεννητικότητα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ε, ρόλο. Όχι μόνο η παραγωγικότητα και κάναμε διάφορες προσωμιώσεις πολιτικών, σύγχρονες προσωμιώσεις για τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη που αφορούν την απασχολησιμότητα, το κόστος του εργατικού δυναμικού ε, και τα κίνητρα που δίνουμε στον να εργάζεται περισσότερο κόσμος. Αυτά και ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ, που απαντήσατε στις ερωτήσεις θέσατε ζητήματα προς προβληματισμών για τα επόμενα έτη. Σύντομα θα αποχαιρετήσουμε τους διερμηνείς, άρα θα τελειώσει και η συνεδρίασή μας. Επαναλαμβάνω, ενδιαφερόμαστε όλος ιδιαιτέρως για αυτές τις πληροφορίες. Θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας τις πληροφορίες, να τις στείλουμε στα μέλη που απουσιάζουν, να μελετήσουμε τις λεπτομέρειες. Είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων. Πρέπει να στρέψουμε το όμα και τους εγκεφάλους μας προς το μέλλον, όπως και εσείς. Σας είμαι θα για αυτό που κάνατε. Ευχαριστώ κυρία Κάφμαν και τον Γιώργο και τους άλλους ευχαριστούμε. Και περιμένουμε και τις διαφάνειες για να τις διανύμουμε, αυτές που παρουσιάσατε. Ευχαριστώ και πάλι. Επόμενη συνεδρίαση. 4 Δεκεμβρίου. Απόγευμα. Από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή σας όρεξη.